Okay, colleagues. Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση με το σημείο 11 σχετικά με την αποστολή της Επιτροπής μας στη Γουινέα. Ο Αρχικός της αποστολής ήταν ο Νόρμπερ ε, Νόιζερ, συμμετείχαν και άλλοι φυσικά. Στόχος ήταν να δούμε αν τα διδάγματα από την ε, κρίση του έμπολα αξιοποιήθηκαν ε, κατάλληλα. Θέλαμε να ξέρουμε αν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν, γιατί επενδύθηκαν στα ε, συστήματα υγείας, ε, επέφεραν ε, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Νόρμπερτ, ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Η αποστολή στη Γουινέα έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου. Πέρα από μένα συμμετείχαν η Μαρία Νόισλ και ο Άνταμ Σένσφελντ. Στόχος ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης του τομέα της υγείας στη Γουινέα μετά την ε, επιδημία έμπολα που ε, τη ζωή σε 2.500 άτομα στην ε, χώρα και περίπου 11.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους ε, στην Δυτική Αφρική. Η ε, ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση στην Δυτική Αφρική ήταν πολύ σημαντική. Ε, διέθεσε συνολικά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 870 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Γουινέα η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επίσης ουσιαστική με κινητοποίηση κονδυλίων από την ΕΚ και το εργαλείο για την ε, σταθερότητα και την ε, ειρήνη από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και από το 10ο και 10ο Ταμείο ε, Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πολλά ζητήματα, συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας και την ομάδα από το Γραφείο Στρατηγικής και Ανάπτυξης και την νέα υπηρεσία, Εθνική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Ε, έγιναν επίσης ε, συναντήσεις ε, με διάφορες ΜΚΟ, με εκπροσώπους του ΠΟΗ και με τον πρόεδρο της, ε, του Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ε, ένα από τα συμπεράσματα της αποστολής ήταν ότι έγινε σημαντική πρόοδος στο τομέα της υγείας στη Γουινέα τα τελευταία δύο χρόνια και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ θετικός για την αντιμετώπιση της επιδημίας του έμπολα και για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Γουινέα. Η επιδημία έμπολα ε, αποκάλυψε τις αδυναμίες, την ευαλωτότητα του συστήματος υγείας, την αδυναμία ανταπόκρισης των υγειονομικών αρχών και την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού. Από την ε, κρίση του έμπολα, από τότε που ξέσπασε, η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα εθνικό σχέδιο υγείας για την περίοδο 2015-2024, του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται να εξελίξει. Ο προϋπολογισμός για την υγεία αυξήθηκε από περίπου 2% το 2018 σε περίπου 8% το 2017 και ε, έγιναν 4.000 προσλήψεις, ε, προσλήψεις 4.000 ατόμων ε, υγειονομικού προσωπικού σε όλη τη χώρα. Υλοποιήθηκε επίσης ε, προληπτική πολιτική κατά των ε, λοιμόξεων και ιδρύθηκε Εθνική Υπηρεσία Γενομικής Ασφάλειας τον Ιούλιο του 2016 με στόχο να ενισχυθεί ε, το σύστημα επιδημιολογικής εποπτείας και να ενισχυθούν οι ικανότητες ανταπόκρισης σε μια ενδεχόμενη επιδημία στο μέλλον. Αντλήσαμε διδάγματα από αυτή τη κρίση ε, συζητήσαμε ανοιχτά με τον Διευθυντή Χώρης του ΠΟΕ σχετικά με τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε να εξέλθει να ανταποκριθεί η διεθνής ε, κοινότητα. Η θετική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας έμπολα ε, τονίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής. Στα πλαίσια του προγράμματος, δύο απογευματινές συνεδριάσεις αφιερώθηκαν στην παρουσίαση των δύο ε, προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το σχέδιο Prepare και το πρόγραμμα PASA. Το πρόγραμμα Prepare χρηματοδοτήθηκε από το περιφερειακό πρόγραμμα του, ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης με κονδύλια 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υλοποιήθηκε από την Expertise France και υποστηρίχτηκε από περιφερειακές ομάδες που είχαν υπό την ευθύνη του την εποπτεία, τον έγκαιρο εντοπισμό και την γρήγορη ανταπόκριση. Με τη διάθεση 29,5 εκατομμύριων ευρώ το πρόγραμμα ΠΑΣΑ συνέβαλε στην ενίσχυση των ικανοτήτων του Υπουργείου Υγείας, στη βελτίωση της λειτουργίας και της χρηματοδότησης της ε, ε μητρικής και παιδικής υγείας και στην υποστήριξη του κεντρικού φαρμακείου της Γουινέας. Ε, επισκεφτήκαμε τις... Ε, το ε, κεντρικό φαρμακείο και το εθνικό εργαστήριο που ελέγχει την παραγωγή φαρμάκων. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στο τομέα της υγείας χρειάζονται ακόμη ε, σημαντικές επενδύσεις Η Γουινέα σήμερα είναι καλύτερη προετοιμασμένη για να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη ε, επιδημιολογική κρίση στο μέλλον. Όμως ε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας μακροπρόθεσμα. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει ε, το σύστημα υγείας στη Γουινέα μέσα από την δημοσιονομική στήριξη. 40 ε, εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για την υγεία στα πλαίσια του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος 2014-2020 και το ε, δεύτερο πρόγραμμα ΠΑΣΑ βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Έχουμε, συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της αποστολής και για τα θέματα της αποχέτευσης και του ε, ακροτηριασμού ε, των ε, γεννητικών οργάνων. Στην Γουινέα έχει υιοθετηθεί νομοθεσία για την απαγόρευση αυτής της πρακτικής. Έχουμε, ε, λάβαμε ενημέρωση από εκπροσώπους του Ταμείου του ΟΗΕ για τον πληθυσμό και από την UNICEF ε, οι δύο αυτοί οι οργανισμοί του ΟΗΕ υλοποιούν ένα κοινό πρόγραμμα στην περιοχή. Και ε, προτεραιότητα στην Γουινέα πρέπει να είναι η κατανομή, σωστή κατανομή του ε, προϋπολογισμού και η ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών. Στην Επιτροπή ΔΕΒΕ πρέπει να συνεχίσει η υγεία να είναι προτεραιότητα και να ασκούμε πίεση για την διάθεση ε, περισσότερων κονδυλίων για την υποστήριξη της υγείας και της εκπαίδευσης ε, στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας καθώς και την ενίσχυση κάθε των παγκοσμίων πρωτοβουλειών και την υγεία. Θα ήθελα εκ μέρους της αποστολής να ευχαριστήσω θερμά την, αποστολή της την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουινέα για την υποστήριξη που λάβαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αποστολής. Όλοι ε, συμμετείχαν και μας βοήθησαν πολύ κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας στη Γουινέα και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουινέα κάνει εξαιρετική δουλειά και μας βοήθησε πάρα πολύ από την αρχή μέχρι το τέλος της αποστολής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Νόρμπερτ. Βλέπουμε λοιπόν πως έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις στον τομέα της υγείας έτσι ώστε να αποτραπεί ε, η νέα εμφάνιση τέτοιου κρούσματος. Ε, πώς θα το αξιολογούσες εσύ. Σε γενικές γραμμές είναι θετικά τα πράγματα, όμως δεν υπάρχουν οι ικανότητες. Έχουν γίνει βελτιώσεις, υπάρχει ευαισθητοποίηση, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις με τις οποίες συναντηθήκαμε ασχολούνται ενεργά με την αντιμετώπιση σίγουρα έχουν αντλήσει διδάγματα, όμως χρειάζεται χρόνος και ακόμα περισσότερο χρήμα. Ο Σαρλ Γκέρντς, ο εισηγητής μας, θα πάρει το λόγο. Και μετά θα μιλήσουμε για τη Σιέρα Λεόνε. Κύριε Γκέρντς, έχετε το λόγο. Μία ερώτηση μόνο. Έχει γίνει κάποια αξιολόγηση όσον αφορά την επιτευθύνσα πρόοδο από την αρχή της κρίσης του έμπολα στη χώρα. Και τι έχει διαπιστώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και για την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση έχει βρεθεί πρόοδος. Για ακόμα πολλά οφείλουμε να κάνουμε. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή σε λίγο, διότι υπάρχουν συστάσεις από τη δική σας έκθεση για τον ε, έμπολα. Μία από αυτές ήταν να ε, υπάρχει εμβολιασμός, ε, να μην ακυρωθεί το όλο πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί κάθε φορά που υπάρχει, υπάρχουν κρούσματα έμπολα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε συμπτωματικά την κατάσταση και μετά επιστρέφουμε στα ίδια. Ε, ο Επίτροπος Αρμόδιος για θέματα υγείας ίσως θα είναι αρμόδιος να απαντήσει. Ε, όμως θέλετε να πείτε για τη Σιέρα Λεόνε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Πώς θέλετε να σας τα πω, αγγλικά ή ισπανικά. Ισπανικά. Α, ισπανικά. είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με αυτό τον φορέα των ιερέων ε, τον επικεφαλής, τον Πορτογάλο ή Βραζιλιάνο που έχουν αυτό τον φορέα λοιπόν ούτως ώστε να βοηθήσουν ανήλικες να τις σώσουν από την πορνεία στην τους καλέσαμε, δεν μπόρεσαν να έρθουν, πάντως υπάρχει ένα βίντεο, και ένα βίντεο το οποίο μπορούμε να το δούμε. Πολύ σκληρό αυτό το βίντεο. Και αφορά αυτές τις ε, κοπέλες, περισσότερες μόνες τους που είναι στο δρόμο. έχουν χτυπηθεί και αυτές από τον ε, ιό. Είναι ηλικία 11 με 17 ετών και κατέφυγαν στην πορνεία γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν και ο μόνος τρόπος να έχουν κάποιον να τις προσέχει, να τις φυλάει τα γνωστά. Και βοήθησαν 200 και υπάρχει μια απέσια σκηνή εκεί με τους ε, τους Κινέζους οι οποίοι δουλεύουν το πρωί και μετά το, το, βράδυ πάνε εκεί πέρα σε κάποιο σκάφος για να τις ε, ε βρούνε και είναι φρικτό αυτό γιατί ε, φανταστείτε ακόμα και αυτές που είναι πόρνες ε, ήταν σε φρικτή κατάσταση. Πολύ σημαντικό. Οπότε εμείς ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές της χώρας και είναι πολλές οι χώρες στην Αφρική όπου πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όπως στη Σχεραλεόνε και στο Σουδάν και ε, σας ζητώ αυτό να συζητηθεί, να διαβαστεί στην Επιτροπή, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο πέραν του βίντεο. Ακριβώς τα πλαίσια ίσως της ε, συζήτησης για την προστασία των ελίκων από την εκμετάλλευση. Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση όσον αφορά την δουλειά και υπάρχει και εκμετάλλευση σε επίπεδο πορνείας. Να το δείτε και να αποφασίσετε. Πάντως είναι θέμα που θα πρέπει να το προωθήσουμε. Γιατί με τη δουλειά μας με τις χώρες ΑΚΕ ε, θα, θα πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ευρώπη ε, είναι, αδιανόητα και πάντως πολλές φορές δεν τα θίγουμε αυτά τα θέματα αλλά σίγουρα θα πρέπει ε, αυτό το οποίο εδώ είναι αυτονόητο δηλαδή η απαγόρευση της περιοδικής πορνείας, της πορνείας ανηλίκων αυτό θα πρέπει να περάσει και σε εκείνες τις χώρες άρα αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε παρακαλώ Ευχαριστούμε πολύ Σίγουρα πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο αυτήν την πρωτοβουλία και γιατί με τον Σαρλ ε, Γκέρντς είδαμε και στην Ουγκάντα για παράδειγμα πολλά κορίτσια ε, χωρίς γονείς, μητέρα, πατέρα για να τα προστατεύσουν και ήταν ευάλωτα στο να πέσουν θύματα. Είναι πάρα πολύ νέες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ θα θέλατε να πάρετε το λόγο. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα κάνετε στον τομέα της υγείας. Να πω ότι σε ό,τι φορά τις ερωτήσεις για την αξιολόγηση, όλα μας τα προγράμματα και τα έργα υποβάλλονται σε ε, ενδιάμεση και μακροπρόθεσμη γενικότερη αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή, στην προκειμένη περίπτωση, ασχολήθηκε με τα προγράμματα καταπολέμησης του έμπολα και τα προγράμματα αυτά ε, χωρίστηκαν σε δύο στάδια, το ΠΑΣΑ 1 και το ΠΑΣΑ 2. Η αξιολόγηση λοιπόν έγινε σε δύο στάδια έτσι ώστε να δούμε τι θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε μετά την εμπειρία μας από το ΠΑΣΑ 1 προτού προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ΠΑΣΑ 2. Επίσης, Πέρα από τη στήριξη των έργων αυτών, προχωράμε σε μία προσέγγιση πιο ε, διαρθρωμένη για τα δημοσιονομικά. Κατανομή πόρων στον τομέα της υγείας. Όπως ε, ακούστηκε, πάμε από πολύ χαμηλά ποσοστά, 2%, ε, και ανεβαίνουμε. Τώρα είμαστε στο 7%. Μετά, ε, σε ό,τι φορά την υλοποίηση, την εκτέλεση του προπολογισμού, που είναι κάτι διαφορετικό, ε, έχουμε και εκεί αύξηση ετήσια. Προσπαθούμε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μια μελλοντική κρίση και να υλοποιούμε διάφορα προγράμματα στη Γουινέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα que está especialmente dedicada a la violencia contra Έχουμε αυτή την πρωτοβουλία για την βία των γυναικών και υπάρχουν κάποια προγράμματα σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο και τέλο πάντων μπορούμε να καταρτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία ε, υπό την αιγίδα για υποστήριξη ως επιτοπλίστων του ΟΗΕ και με τη συνεργασία διαφόρων διεθνών φορέων σε κάποιες χώρες. Δεν το έχουμε εξειδικεύσει ένα χώρα, είναι μια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί ε, για χρήση σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλος από την Επιτροπή. Α, από την ΕΚΟ. Όχι. Είμαι από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Απλώ να σα ευχαριστήσω θερμά. Και έχουμε τα δύο θετικά για την ε, τεύματα πρόοδου στην ε, Γουινέα αλλά και την ε, πρόοδο όσον αφορά τον ιό έμπολα. Σημαντική βοήθεια του ΟΗΕ. Θετικό, θετική πρωτοβουλία σποντά. Όπως αναφέρθηκε αντιμετωπίζεται έτσι και το θέμα των γενετησιών ακροτηριασμών. Στον Κογκό τώρα ναι έχουμε ξέσπασμα αυτής της ε, ασθένειας του έμπολα. και δεν ξέρω πώ τώρα ξέρουμε περισσότερα που επεμβαίνουμε ε, κατεπηγόντω παρά τον είχαμε βοηθήσει να στηθεί ένα σύστημα υγεία. Να δούμε τι γίνεται με την έκθεση Γκέρενς εκεί στα συμπεράσματα, να δούμε τι θα πρέπει να προωθήσουν προς την πλευρά της Επιτροπής για τα θέματα των εμβολίων. Σας θα πούμε και στον Επίτροπο. Εδώ και τρία έχει ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία στη συνεργασία με τον Αντρέο Κάτης και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και δυστυχώς υπάρχει αυτό το κλασικό σχήμα του να γίνονται μαζικές προσπάθειες και έρευνα για κανένα τρίμηνο εξάμεινο όσο έχει δημοσία το θέμα και μετά να σβήνει η προσπάθεια. Άλλο. Κύριε Σνόιζερ, να προσθέσω και κάποια προσωπικά σχόλια. Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προορατικοί. Μόνο έτσι θα κάνουμε σωστή δουλειά. Τα διδάγματα που αντλήσαμε από την περίπτωση του έμπολα, όχι μόνο εμείς αλλά και η ίδια η χώρα, θα μας βοηθήσουν στο μέλλον να εφαρμόσουμε πολιτικές. Δυστυχώς θεωρούμε πως αυτή η εφαρμογή ε, καθυστερεί και γίνεται με πολύ αργούς ε, ρυθμούς. Όμως, στον προϋπολογισμό βλέπουμε τετραπλασιασμό των ε, κονδυλίων για την υγεία. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Γι' αυτό μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε δημοσιονομικά ε, τη χώρα εφόσον έχει βελτιωθεί και η δομή. 4.000 επιπλέον επαγγελματίες υγείας είναι καλά νέα, είναι μια καλή απάντηση, όμως ε, η κατάρτιση νέων ε, γιατρών και λοιπόν επαγγελματιών υγείας ε, είναι χρονοβόρα. Μαζί όμως με την τεχνογνωσία των Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων νομίζω πως πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, για το θέμα της αξιολόγησης ο Σάρλ έχει δίκιο. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον Μπόι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημάνουμε και να πετήσουμε. Επίσης, πρόοδος έχει σημειωθεί και σε ό,τι φορά τη διανομή φαρμάκων. Αυτό είναι ένας τρόπος ε, γρήγορης και Κατάλληλη αντίδραση όταν υπάρχει ένα ξέσπασμα κρουσμάτων έμπολα. Όμως δεν αρκεί σε περίπτωση επιδημίας. Για παράδειγμα, σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει σε κεντρικό επίπεδο διακυβέρνησης να υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, τα οχήματα για παράδειγμα, που θα διανύμουν τα φάρμακα σε όλες τις περιοχές που έχουν σημειωθεί κρούσματα. Μετά υπάρχει και το θέμα των νέων οι οποίοι ε, πάσχουν, ασθενούν από έμπολα. Υπάρχει μετά ε, κοινωνικό στίγμα, κοινωνικός αποκλεισμός των ανθρώπων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως θα πρέπει να αναλάβουμε δράση έτσι ώστε να ε, προωθήσουμε την ένταξη ή την επανένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία. Επιπλέον, να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μαστίζεται από ένα τεράστιο πρόβλημα απορριμμάτων. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά σκουπίδια σε μια χώρα. Μάλιστα υπάρχουν ολόκληρες πόλεις όπου οι κάτοικοι ζουν μέσα στα σκουπίδια. Είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν ε, υπάρξει κάποιες αρχικές δράσεις, όμως ε, δεν θα πρέπει να σας εκπλήσει το γεγονός ότι ξεσπάνε ε, ε, τέτοια κρούσματα έμπολα και δεν είναι απίθανο να ξεσπάσει και επιδημία όταν υπάρχει τέτοιο υγειονομικό πρόβλημα. Αυτή είναι μια υγειονομική βόμβα διότι πρόκειται για θανάτους από έμπολα 10, 12 και παραπάνω ατόμων οι οποίοι ζούσαν μέσα στα σκουπίδια. Χρειάζεται λοιπόν άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος ε, των ε, απορριμμάτων, της ε, διαχείρισης αυτών. Είναι αυτό όμως και τμήμα των υγειονομικών δράσεων που θα πρέπει να αναλυφθούν. Τέλος, η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία και η Γουινέα, όλη αυτή η περιοχή νομίζω πως ε, έχει και κάτι θετικό. Χαρακτηρίζεται από σχετικά σταθερές ε, κυβερνήσεις, πολιτική σταθερότητα. Στη Γουινέα υπάρχει μια σχετικά σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει καλές επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δομές ε, του κράτους είναι σχετικά σταθερές. Μετά στη Σιέρα Λεόνε ε, έχει υπάρξει μια αλλαγή ε, εξουσίας και, θεω... και στη Λιβερία το ίδιο. Θεωρώ λοιπόν ότι όσο σταθεροποιείται ακόμα περισσότερη κατάσταση θα βελτιωθεί και το πρόβλημα ε, το υγειονομικό. Ευχαριστώ πολύ Νόρμπερτ. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς. Πρέπει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση και να φροντίζουμε να ελέγχουμε ότι τα χρήματα πηγαίνουν πραγματικά στον τομέα της υγείας. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα σε λίγο. Περιμένουμε τον Επίτροπο. Um, Καλησπέρα σας και πάλι συνάδελφοι. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 12, ένα πολύ σημαντικό σημείο. Πρόκειται για το διαρθρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος. Παρότι του χρόνου θα υπάρχει νέο πρόγραμμα εργασίας, Νομίζω πως ε, κανείς μας δεν πιστεύει, κύριε Πίτροπε, ότι φέτος είναι το τελευταίο, η τελευταία πλήρης χρονιά κοινοβουλευτικής ε, θητείας, αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Πριν, πριν έρθετε συζητούσαμε την κρίση με τον ιό του έμπολα. Ο Νόρμπερτ Νόιζερ είχε πάει με μια αποστολή στη Γουινέα Γι' αυτό λοιπόν ε, τρία χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που συζητήσαμε μαζί εδώ αυτό το θέμα και νομίζω πως πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με τον Επίτροπο κύριο Στυλιανίδη για τα ε, πολύ σημαντικά ε, κρεμή ζητήματα. Για μας είναι η εκπαίδευση των παιδιών, η περιπτώση έκτακτης ανάγκης και ε, όλος ο σύνδεσμος μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας, χρηματοδότησης, έργων και αποτελεσμάτων. Στην Ουγκάντα είδαμε με τα μάτια μας κάποια από τα προβλήματα που έχουν προκύψει ε, σχετικά με την χρηματοδότηση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά εκκρεμή ζητήματα από το παρελθόν, αλλά βέβαια και τον ε, Ιούνιο θα έχουμε νέα προγράμματα. Το νέο, η νέα πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, νέο τήσιο πρόγραμμα για την αναπτυξιακή πολιτική, δεν γνωρίζω αν θα έχουμε και νέο πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά ε, είναι πολλά στο πρόγραμμα για τον Ιούνιο. Να πω επίσης στους συναδέλφους μου ότι μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Επίτροπο Στυλιανίδη και αύριο με τον Επίτροπο Μίμητσα, η Επιτροπή μας θα συντάξει μια πρόταση που θα απαριθμεί τις προτεραιότητές τη για το επόμενο έτος, θα τη στείλει στη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών και αυτό θα οδηγήσει σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προσδοκίε μας για τα επόμενα έτη. Κύριε Στυλιανίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Λίντα, αγαπητοί συνάδελφοι. Και σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου σήμερα να είμαστε μαζί. Και γνωρίζετε ότι αυτό ο δομημένο, διαρθρωμένο διάλογο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψει για ε, τις ε, προτεραιότητες, για τα λειτουργικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και για τη διαχείριση των ε, κρίσεων αυτά δηλαδή που έχει το χαρτοφυλάκιό μου. Οπότε, όπως ξέρετε, οι συμβουλές σας, η συνεργασία σας, η βοήθειά σας ήταν ανεκτήμητα για αυτήν την ε, τετραετία και σας ευχαριστώ ε, όσον αφορά την συνεργασία μας στην Άριστη. Επίσης υπάρχει κι άλλος ένας ε, λόγος για να προβώ αυτές τις διαπιστώσεις. Τώρα σε αυτόν τον τελευταίο διευθυνμένο διάλογο μου έχετε ζητήσει να έχουμε ένα έγγραφο για τα και κάτι το οποίο είναι κορυφή προτεραιότητα ήδη τα ανέφερε η Λίντα και μπορούσα να πω ότι πρόκειται για κάποια πραγματική μου αιμονή που όμως έχει τη θετική πλευρά και σήμερα με μεγάλη μου χαρά μπορώ να σας πω ότι τηρούμε τα όσα έχουμε τάξει και υποσχεθεί ε, σε εσάς γιατί πρόκειται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ε, εγκρίνει αυτό το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο θα έχουμε τις άριστες πρακτικές και στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε μόχλευση για περισσότερους πόρους, να αναβαθμίσουμε την συνεργασία και να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια μορφή, να διαμορφώσουμε δηλαδή το όλο θεματολόγιο τα τελευταία 34 χρόνια έχουμε γίνει πρωτοπόροι σε παγκόσμιο ελληνικές όσον αφορά τι κατεπίγουσε καταστάσει. και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μα στηρίξατε πολιτικά και δημοσιονομικά και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνση για την ανθρωπιστική δράση ΕΚΟ αλλά και τις αντιπροσωπείες μας ε, και πάλι σας ευχαριστώ. Άλλη μια εξέλιξη θετική. Πρέπει να την αναδείξουμε όσον αφορά δηλαδή την χρηματοδότηση. Μια που Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μόλις έκανε τις προτάσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία χάνεται ένας ε, μέγας πληρωτής όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά θα πρέπει η απογοήτευσή μας ε, να ειδωθεί σαν μια ευκαιρία και να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε συγκεκριμένη ανταπόκριση στα προβλήματα του μέλλοντος και στις προκλήσεις θα πρέπει να γίνουν βέβαια περικοπές δαπανών σε κάποιους τομείς το δυστυχώς είναι αναπόφευκτο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε κατά νου το τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να στείλει ένα θετικό μήνυμα. Οπότε κάνουμε 30% αύξηση στον ανθρωπιστικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι εντελώς απαραίτητο. Γνωρίζετε καλά ότι οι ανάγκες με τη μέρα αυξάνονται. Η βοήθειά σας θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Πιστεύω ότι η αύξηση του 30% είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ιδίω για την περίοδο μετά την αποχώρηση της ε, Βρετανίας. Κάτι άλλο θετικό. Για την πολιτική προστασία προτείνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη αύξηση, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, θεομηνίες για τις φυσικές καταστροφές σε ενωσιακό επίπεδο και επίσης να δούμε το, για το πώς θα αναβαθμίσουμε τη δυνατότητά μας ανταπόκρισης για ένα σωρό δύσκολα προβλήματα. Και λόγω των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος αυτές οι περιπτώσεις εντυπωσιακά αυξήθηκαν. Συνάδελφοι, τρία θετικά μηνύματα όσον αφορά τους κοινούς μας στόχους, ευθύνες και νομίζω ότι φέτος μπορούμε με ενθουσιασμό να στόχουμε στη δουλειά ούτως ώστε να επιλύσουμε όχι μόνο τα κλασικά προβλήματα αλλά και ένα σωρό δυσάρεστες εκπλήξεις που αντιμετωπίζουμε. Θα δούμε τώρα κάποιο άλλου είδους ε, λειτουργικά πιεζιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εφαρμογή της πολιτικής μας. Δυστυχώ. οι ανθρωπιστικές ανάγκες τελευταίο χρόνο δεν έχουν μειωθεί. Μέρα με τη μέρα οι ανάγκες αυξάνονται. Θέλω να αρχίσω από το έργο μας στην Μέση Ανατολή που είναι στην γειτονιά μας. Αλλά από την άλλη μεριά είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των πιο δραματικών εξελίξεων της επικαιρότητας και βέβαια θα πρέπει αυτό ε, αναπόφευκτα να το αντιμετωπίσουμε. Είναι καθήκον μας, ηθική μας υποχρέωση να προσέξουμε τι γίνεται εκεί. Η Συρία μπήκε στην 8η χρονιά εμφυλίου. 13 εκατομμύρια είναι οι Σύριοι που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα για την προστασία, την ε, προσβασιμότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι καταβάλουν προσπάθειες όσον αφορά κάποιες ε, πολιορκικούμενες περιοχές, θέματα ασφαλείας και Επίσης έχουν μισό τους κινδύνους για όσους ε, ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια και να μπορούν αυτοί έγκυρα να προσφέρουν την ε, αρρωγή, την ανθρωπιστική. Ο πόλεμος στην Συρία έχει γίνει αιτία για ε, εκτοπισμό προσώπων για πάρα πολλούς πρόσφυγες και στην Τουρκία και στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Πολλέ φορέ αυτά είναι σε μεγέθη δυσανάλογα για τον πληθυσμό της χώρα. Όπω γνωρίζετε, στον Λίβανο έχουμε 40% του πληθυσμού που είναι πρόσφυγες. Μπορείτε να το φανταστείτε. Σκεφτείτε να υπάρχει τόσο υψηλό αριθμό προσφύγων σε αυτή την τόσο ευάλωτη χώρα που έχει και τόσο ευμετάβολο ε, πολιτικό σκηνικό. Βέβαια, τι τελευταίε εβδομάδε γίνανε εκλογέ που έστειλαν θετικό μήνυμα. Επίση, να μην παρέψουμε να πούμε τις προσπάθειές μας για το ESSM. Υπάρχει αυτού του είδους το δίκτυο ασφαλείας όσον αφορά τη διαμετακόμιση των προσφύγων ε, διαμέσου της ε, Τουρκίας. Στην Τουρκία φιλούσαν 3,8 εκατομμύρια μεταναστών και καλύπτουμε με την βοήθειά μας 1,3 εκατομμύρια. Είναι το πιο μεγάλο μας ανθρωπιστικό πρόγραμμα που έχουμε ποτέ εφαρμόσει. Επίσης, επανελειμμένα επισκεφτικά τη χώρα για να δω πώς πάνε εκεί οι προσπαθειές μας, να δω τι ισχύει επί τόπου και ένιωσα υπερήφανος για το πρόγραμμα μας. Μια που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την βοήθεια προς τους ε, πρόσφυγες για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια για να ξεβρεθούν τρόποι ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε την τοπική κοινότητα με τους πρόσφυγες. Βέβαια και το e ΙΕΣΕΣ έμεινε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο έχει σχέση με την παιδεία. Και γνωρίζετε πριν από λίγους, ε, λίγες οργανώσαμε την ε, δεύτερη διάσκεψη για την Συρία στις Βρυξέλλες και κινητοποίησαμε 6,2 δις ευρώ. Η Ένωση και τα κρατημέλη και πάλι ήταν οι πιο μεγάλοι δωρητές. Με 7% καλύψαμε από όλη αυτή την ανθρωπιστική προσπάθεια. Άρα εμείς είμαστε ο πιο μεγάλος δωρητής όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης της Συρίας. Δυστυχώ όμως αυτό είναι ένα μόνο από τα προβλήματα αυτής της περιοχής στην Ιεμένη. Ε, Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι σοπεδοτικές για αυτή την έτσι γαλλιώς ευάλωτη και φτωχή χώρα σχεδόν 75% των γεμενιτών χρειάζονται βοήθεια. Προσπαθήστε να φανταστείτε ποια είναι η κλίμακα, ποιο είναι το μέγεθος των αναγκών. Και Είχαμε ένα γεύμα εργασίας με τον Γενικό Ραμβλίο του ΓΕΙ, τον κύριο Γκουτέρε, και αναφερθήκαμε και στο Συριακό αλλά και στην Ιεμένη ε, και είπε κάτι θετικό. Είπε ότι θα έχουμε νέο κύμα διαπραγματεύσεων ε, μεταξύ των εμπλεκομένων. Ενώ στην προσευχή γιατί στην Ιεμένη πολλές φορές η κατάσταση οδηγεί σε προβολές επόδυνες εκπλήξεις. Πάντως, το περασμένο μήνα είχαμε την διάσκεψη για την Ιεμένη και τα κράτη-μέλη για άλλη μια φορά έδειξαν ότι χαρακτηριζόμαστε από αλληλεγγύη και ανθρωπιά προς ε, τους γεμενίτες. Και όλοι μαζί εισφέραμε 500 εκατομμύρια δολάρια είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό κομμάτι τη όλης πρικοδότηση. Οι ανθρωπιστικέ συνέπειε, κυρίε και κύριοι, από όλου αυτού τους πολέμου στη Μέση Ανατολή, ε, μας φύγουν άμεσα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. ότι στην Ευρώπη τα θεσμικά όργανα ειδικότερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Όμως ιδίω όσον αφορά το προσφυγικό ε, η κατάσταση έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις ε, ιδίω στην Ελλάδα υπάρχει άλλωστε και ο διάδρομος των μεταναστών και προσπαθούμε να προσφέρουμε αρρωγή μέσα στα βαθιά σύνορα οπότε θα πρέπει και πάλι να σας ευχαριστήσω γιατί λόγω ημών καταφέραμε να θεσπιστεί νέα νομοθεσία με μια προσέγγιση ε, σύντομη για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή στην Ελλάδα. Ξαναπήγα στη χώρα την περασμένη εβδομάδα. Πραγματικά κάθε φορά που πάω βλέπω βελτίωση των συνδικών εκεί επιτόπου, ιδίως ε, όσον αφορά την υπηρετική χώρα. Άρα το ότι έχουμε κάποια ε, νησιά του Αγίου, ιδίω στην Λέσβο, που το πρόβλημα έχει δημιουργήσει επώδυνε συνέπειε. Και σε επαφή με τι ελληνικέ αρχέ και την κυβέρνηση προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας, ιδίω για τα νησιά του Αιγαίου. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αύξηση των αφήξεων ιδίως μέσω του διαδρόμου του Εύρου. Τα είπαμε επίση και με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βίτσα. Φτυχώς ε, η κατάσταση βελτιώθηκε, ήδη μειώθηκαν οι αυξήσει. Πάντω θα πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού για να δούμε τι θα κάνουμε με οτιδήποτε νέε αφήξει. Πάντως διατηρώ την αισιοδοξία μου για την κατάσταση στην Ελλάδα, ιδίω όσον αφορά την υπηρετική χώρα. Γιατί έχουμε και ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Εστία, που είναι πάρα πολύ καλό. Με αυτό το πρόγραμμα μπορέσαμε να προσφέρουμε στέγη στους ε, πρόσφυγες και ήδη έχουμε καλύψει 35.000 προσφύγων. Το Ιράκ Συνεχίζουμε να βοηθούμε τη χώρα. που έδωσε και κέρδισε την μάχη κατά της βίας, της τρομοκρατίας, του μίσους, του Ισλαμικού κράτους. πολλές φορές και εσείς και εμείς εμείναμε σε τέτοια προσέγγιση ότι θα πρέπει δηλαδή να συνεχιστούν οι προσπαθίες μας ούτω ώστε να νικήσουμε το Ισλαμικό κράτος σε επίπεδο ιδεολογίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι εύκολο και την Κυριακή που πέρασε είχαμε δημοκρατικές εκλογές που ελπίζω ότι θα αποτελέσουν νέα αρχή για τη χώρα. Πρόκειται για μια καινούργια αρχή. Να δούμε. Στο Ιράκ έχουμε εισφέρει 350 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 και για το 2018 θα δώσουμε κι άλλα. Τώρα να δούμε και τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Συνεχίζουμε το ανθρωπιστικό μας έργο στην Παλαιστίνη σε επαφή με τον Γενικό Γραμματείο του ΟΗΕ ενεργούμε εμπιστευτικά και η περισσότερη βοήθειά μας πάει μέσω των διάβλων της Digineer συντριπτική πλειοψηφία των στοιχείων βοήθειας και επίσης έχουμε ανθρωπιστεί και αρρωγή μέσω της Γενικής Διευθύνσης ΕΚΟ και ανεβήκαμε στα 24 εκατομμύρια ευρώ για το 2018 επίσης και στη συνεργασία με τους φορείς και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Να μπορούσαμε να καλύψουμε τις πιο επίγουσες ανάγκες στην Παλαιστίνη. Όμως, αυτό με ανησυχεί περισσότερο είναι το ότι έχει ενταθεί τώρα στις μέρες μας η βία στην Γάζα. Ε, επίσης, έχουμε ε, ιδιαίτερα πολλούς και τραγικούς θάνατους και άνω της βίας λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ δίνηρο και η κατάσταση ήταν που ήταν ε, κακή έχει γίνει τώρα χειρότερη και εύκολα μπορούμε όλοι μας να αντιληφθούμε τη λόγω αυτών των τελευταίων εξελίξεων η κατάσταση χειροτερεύει μέρα προς μέρα. Μιλούμε για μια παγκόσμια πλέον απειλή. Και όπως αναφέρθηκε από την υπάτη εκπρόσωπο στην τελευταία της δήλωση, το Ισραήλ θα πρέπει να αποστεί από δυσανάλογη και υπερβάλλουσα χρήση βίας. Πάρα πολύ σημαντική νομίζω η δήλωσή της. Αλλά ε, η Χαμάς θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι διαδηλώσεις δεν θα έχουν βίο χαρακτήρα. Ισορροπημένη η δήλωση αυτή της υπάρξης εκπροσώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να έχει αυτόν τον σημαντικό ρόλο της και να μπορέσει να είναι επικοδομητικός συνομιλητής. Ιδίω μετά τις εξελίξει. εξελίξεις. Ε, πήγα στο Κονγκό για να δούμε λίγο την Αφρική τον ε, Μαρτίο. Ξεκίνησα από το νοσοκομείο Μπάτζι. Ήρθα σε επαφή με τον φίλο τώρα, Μουγκέγια τον βραβευμένο και με συνεκλώνησε, με συνεκίνησε η δουλειά του εκεί. Ήταν βεβαιοδυνηρή αυτή η εμπειρία που ε, συνάντησα τόσες ε, περιπτώσεις, τόσες γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Επίσης, ε, ένιωσα περήφανος για τις επιπτώσεις της βοήθειάς μας Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε μέρα έτσι σώζει ζωές. Και εσείς είχατε πάει στον Σομίτς, δεν είναι στον Πάντζ, ναι, ναι, λέει ο Πρόεδρος. Επίση στην Κινσάς έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση για το ποια είναι τα προβλήματα Στην Γενέβη είχαμε αυτή τη διάσκεψη την πρώτη για το Κονγκό για να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες. Δεν συμμετέσχει η κυβέρνηση. Ε, μαζέψαμε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, μεγάλο κατόρθωμα. Ε, μεγάλο κατόρθωμα γιατί μέχρι πριν από λίγο ήταν μια κρίση ξεχασμένη. Και μαζί με το μπάτζι ε, πρόκειται για επιτεύγματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η συμμετοχή μας, η συμβολή μας ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό σε σχέση με τις παγκόσμιες ανθρωπιστικές προσπάθειες. Τώρα να μιλήσουμε και για την πρόσφατο ξέσπασμα του έμπολα στο Κονγκό. Παρακολουθούμε από κοντά τις εξέλιξεις και έχω τη επαφή με τον Γενικό διευθυντή από τον ΠΟΕ. Μίλησαμε μόλις χθες και είμαστε έτοιμοι να πάμε για να βοηθήσουμε κατεπηγόντως με τον Ευρωπαϊκό Φορέα ε, Γιατρών που έχει η Ένωση. Θα πρέπει ποτέ να εφησυχάζουμε όσον αφορά τον έμπολα και ασχολούμαι και σε επίπεδο συντονισμού με αυτό. Και όπως είπαμε και με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Υγείας η κατάσταση είναι υπό έλεγχο μέχρι σήμερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταθέσουμε τα όπλα. Να φυσικάσουμε επίσης για το κέρα της Αφρικής, εκεί συνεχίζεται η ξηρασία, 13 εκατομμύρια χρειάζονται βοήθεια, φαΐ, φαΐ επίσης σε Σομαλία, Αιθιοπία και Κένια στο Νότιο Σουδάν συνεχίζεται ο εμφύλιος και γνωρίζετε ότι έχω αποκρισταλωμένες θέσεις για το Σουδάν, ότι πρόκειται για μια ντροπή. Η κατάσταση εκεί είναι τόσο δύσκολη που εκατομμύρια, εκατομμύρια ε, εξαρτώνται 100% από την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά την Αφρικανική δημοκρατία, μερικοί από εσά πήγατε στα τα μέσα Φεβρουαρίου με αποστολή εκεί και είδατε τη σκληρή πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα. σε διάφορου επισήμου εδώ και διαπιστώσαμε από κοινού ότι είναι βασικό θέμα το να επικρατήσει ασφάλεια Πρόκειται για μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και βέβαια για αυτή την κρίση ε, έχουμε πάρα πολύ λίγα κονδύλια. Εκτιμώ το ότι εσείς πήγατε και διατρανώσατε το ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα προς ότι προσπαθούμε ότι σε επαφή με ε, την κυβέρνηση και με τις υπηρεσίες ασφαλείας ε, γίνεται προσπάθεια για να βρεθούν καλύτερες ημερομηνίες για το Σαχέλ τώρα. Ε, το Σαχέλ συνέχεια βρίσκεται σε κρίση. Πόλεμος, ε, αλλαγή του κλίματος, όλα αυτά φρενάρουν την πορεία προς την ειρήνη και την ευημερία. Δεν είναι δυνατόν όμως να έχουμε εδώ μια κρίση ξεχασμένη. Το τι θα κάνουμε γενικώ με την Αφρική θα καθίσει το μέλλον των επόμενων γενιών ε, και για την Αφρική αλλά και για την Ευρώπη. θα γνωρίζετε ότι πάρα πολλές ροές προσώπων γίνονται προς την Ευρώπη. Ασία. πρόκειται για μια ανθρωπιστική τραγωδία, τι έχει γίνει με τους ε, πρόσφυγες ε, Ροχίγκα και πήγα στο Μιανμάρ, πήγα στο Μπαγκλαντές τον Οκτώβριο του 2017, επισκέφθηκα το παζάρι στο Κόξ, είδα εκεί πέρα κάτι το οποίο με σόκαρε, γιατί εκεί έχουμε 600.000 πρόσφυγες που στριμώχνονται ε, και προσπαθούν να επιζήσουν σε μια έκταση 13-14 ε, τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ε, συνεχίζεται επομένως, η έξοδος προς Μαλαισία και Μπαγκλαντές. Και η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης Μπαγκλαντές και της κυβέρνησης των Μιανμάρ για τους Ροχίνγκα, η συμφωνία δεν εφαρμόζεται. Και οι συνθήκες για επιστροφή δεν υπάρχουν. Οπότε όλες αυτές οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πάντως εμείς συνεχίζουμε να βοηθούμε. Για μας είναι ηθική επιταγή. Τέλος. Να σας πω δύο λόγια για την αποστολή στην Νότιο Αμερική τον Μάρτιο. Πήγα στην Κολομβία, και συνεχάρην τον Πρόεδρο Σάντος για το θάρρος, την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει την πορεία προς ε, συμφιλίωση και ε, την ειρήνη. Ξέρω και από τη δική μου πατρίδα πόσο δύσκολη υπόθεση είναι η εθνική συμφιλίωση, πόσο μακρά η διαδρομή είναι και τον συνεχάρηκε και για τις επιτόπου προσπάθειες που έχει καταβάλει. Βέβαια όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις ε, στο μέλλον και γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και είδω ότι είναι πολύτιμη η προσπαθία μας σε κάποιες κοινότητες που έχουν φυγεί από την βία στην Κολομβία. Πήγα και επισκέφθηκα τα σύνορα με την Βενεζουέλα και είδα πώς η κρίση στην ε, Βενεζουέλα έχει μεταδοθεί και ε, ε, στην Κολομβία όσον αφορά την δημοσιογή όσον αφορά το, το, το, το, τα είδη διατροφής είναι, που έχουν φυγεί πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Κάποιες γυναίκες πάνε από το Καράκας εκεί για να μπορέσουν να βρουν ένα εμβόλιο για το νεογέννητό τους. Και είδα και άλλες γυναίκες που περπάτησαν, ε, ταξίδεψαν χιλιόμετρα τέλος πάντων, για να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους για να βρουν ε, φάρμακα. πρώτη για ιστορίες πάρα πολύ στενάχωρες. Και είναι πάρα πολλές τέτοιες οι περιπτώσεις και κατά την αποστολή ανακοίνωσα ότι θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση για τα προγράμματά μας. Και όχι μόνο στην ε, Κολομβία, αλλά και στο ιστορικό της Βενεζουέλας με τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε ήρθαμε αντιμέτωποι με συγκρούσεις και με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές αυτό ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι διαπραγματευτικό χαρτί στις περιοχές όπου γίνονται αυτές οι ενοπλές συγκρούσεις. Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι οι στόχοι και έχασαν τη, τη ζωή τους ε, δικοί μας άνθρωποι προσπαθώντας να σώσουν ζωές. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα λοιπόν, ανθρωπιστική κρίση και δημιουργείται και μια ανθρωπιστική κενή ζώνη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι και πρέπει να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Για μένα είναι θέμα αρχής. Χρειάζεται να απαιτήσουμε την ε, συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για όλους, ανεξαιρέτως. Είναι προτεραιότητα όλων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που εδώ στην Επιτροπή σας έχουμε όλοι πάνω κάτω την ίδια άποψη. Όλοι μας είμαστε υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού δικαίου. Έπειτα, η έμφυλη βία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι δυστυχώς πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκή, λοιπόν η ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία και η ενημέρωση για το τι καθιστά έμφυλη βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι πρωτοπόρος στις δράσεις αυτές και στο πλαίσιο των ε, Ευρωπαϊκών ημερών ανάπτυξης θα διοργανωθεί και ένα πάνελ για το θέμα αυτό και θα χαρούμε πολύ διότι στο πάνελ αυτό θα συμμετέχει και η πρόεδρό σας η Λίντα Μακάβαν. Τώρα, να σας πω δύο λόγια για τον δεύτερο πυλώνα των ε, αρμοδιοτήτων μου, την πολιτική προστασία. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πολύ δημιουργική προσέγγιση που είχατε στις ε, περιπτώσεις ε, διάσωσης. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για την έκθεσή του, κ. Ζόφκοφ. Σίγουρα είναι πολιτικό το θέμα. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρότερη Ευρώπης που θα προστατεύει, που θα σώζει ζωές και θα βασίζεται στις αρχές της ε, αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Ίσως θυμάστε τον περασμένο Οκτώβριο μετά την υπόθεση στην Πορτογαλία ο πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε ότι θέλουμε η Ευρώπη να κάνει πολλά παραπάνω από το να εκφράζει απλά συλληπιτήρια. Αυτό είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα και οι συνθήκες μας έδειξαν ότι δεν αρκούν ε, αυτά που κάνουμε προς το παρόν. Το εφιστάμενο σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και να πω εδώ ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με το Γενικό Γραμματέα για την κλιματική αλλαγή. Το πόρισμα είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας όχι μόνο εκτός Ευρώπης, για να πείσουμε δηλαδή τους πολίτες, αλλά και εντός, στα ίδια τα κράτη-μέλη. Οι διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με θέματα διάσωσης έχουν προχωρήσει και εδώ να σας ευχαριστήσω γιατί χάρη σε εσά προχωρά πολύ γρήγορα το θέμα. Και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν γρήγορα, γιατί η επόμενη καταστροφή μας περιμένει στη γωνία, αγαπητοί συνάδελφοι, κυριολεκτικά. Ακριβώς διότι υπάρχει πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγή. Έχω συζητήσει με αρκετούς επιστήμονες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή. και δυστυχώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ε, πιστεύουμε. Όμως, επιτρέψτε μου να βάλω μια τελεία εδώ να πω ότι όπως πάντα είμαι στη διάθεσή σας, είμαι εδώ έτοιμος να ακούσω τις ε, προτάσεις και τις ιδέες σας, διότι όχι μόνο βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι, αλλά ε, έχουμε πολύ περισσότερα που μας ενώνουν από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Επίτροπε. κάθε φορά που έρχεστε, κάθε φορά που έρχεστε και μάλιστα από τότε που γίνατε επίτροπο, τα προβλήματα αυξάνονται. Όχι εξαιτία σα, φυσικά, αλλά εξαιτία των ε, συγκυριών. Σήμερα το πρωί συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών που μας μίλησαν για την κατάσταση στο Σουδάν, όχι μόνο στο Νότιο Σουδάν, αλλά και ε, στο Σουδάν και είδαμε ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Κάθε φορά βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί, όμως πρέπει αυτό να γενικευθεί. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ και μετά έχω έναν μεγάλο κατάλογο μιλητών που ζήτησαν το λόγο. Ενρίκε, έχετε το λόγο ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Χρήστο. Μια με την αλήθεια στην αρχή των όσων μα είπε, έλεγε ότι ο διαδρομένος ε, διάλογος τη επιτροπή μας με εσένα που είσαι ε, ε, εκπρόσωπο τη Επιτροπής πάντοτε είναι κάτι το θετικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει κοινού αγώνες. Σε μερικές περιπτώσεις είχαμε ε, κάποιες επιτυχίες καταπληκτικές όπως η αύξηση της προκοδότησης για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πάντοτε λέμε όποτε συνδυόμαστε ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης κατά κάποιο τρόπο ε, εξορισμού ε, είναι παράγον βοήθειας προς τον Επίτροπο. Και θα πρέπει επίσης να σε ευχαριστήσω γιατί ανέφερε την κατάσταση στην Γάζα, την Παλαιστίνη, την Μέση Ανατολή. Έχουμε αναλάβει προσπάθειες εδώ και πολύ καιρό να μπορούμε να προστατεύσουμε, να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο είδους ε, ευκαιρίες, ευκαιρίες για ανθρωπιστική βοήθεια προς ε, έναν κόσμο που ζει σε μια ε, φυλακή ανθρωπιστικής κρίσης. Κάτι το οποίο είναι ήδη φυλακής επομένως, τους κρατάει και συνεχώς έχουμε το σαμποτάρισμα των όσων δημιουργούμε ως ε, διευκολύνσεις στην Γάζα. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και πολιτικά να βοηθήσουμε και τελικά να υπάρξει κάποιο είδους φρένο, τροχοπέδι στις δραστηριότητες του Ισραήλ. Και είπα έκαναν κάτι σαν αυτό που έκανε ο Αριέλ Σαρών για να ξεκινήσει αυτή η, η κρίση τότε με το μεγάλο τζαμί που τα όσα έκανε ο Σαρών για αυτό το τζαμί οδήγησαν στην ε, δεύτερη Ιντιφάντα και οδηγηθήκαμε σε χιλιάδες ε, νεκρών. Μια τραγωδία που έπληξε και τους Ισραηλινούς. Ε, και πρόκειται για τραγωδία πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Γάζας. Και η Λίντα και εσείς κύριε Πίτροπε αναφερθήκατε και στην κρίση του έμπολα. Ήταν η πρώτη συγκεκριμένη κρίση που θα έπρεπε ως Επίτροπος να αντιμετωπίσετε. Τώρα δεν βλέπουμε ότι υπάρχει νέο ξέσπασμα αυτής της κρίσης και άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που να είναι σταθερό, δομημένο, να έχουμε ένα σύστημα ταχείας ε, αντίδρασης για τέτοιες ε, κρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικός ο ρόλος της παιδείας για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους ε, τραγωδιών. Οπότε όλα αυτά τα οποία ε, έχουμε κάνει σε αυτό το επίπεδο όσα περιέχει σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν είναι πρόληψη τέτοιων κρίσεων. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει γνώσεις στον κόσμο ούτως ώστε να αποφεύγουν μια συμπεριφορά που αποδεικνύεται επικίνδυνη και ε, να αποφύγουν συμπεριφορές που δίνουν μια συνέχεια και διεύρυνση στην ε, κρίση. Επίσης η Ένωση θα πρέπει τώρα να δούμε ε, πού θα καταλήξει για αυτή την αξιολόγηση όσον αφορά την τετραετία ανθρωπική βοήθεια. Να κάνουμε αξιολόγηση, αν θα κάνουμε στο μέλλον. Το Κοινοβούλιο είναι γνωστό ότι έχει εγκρίνει ένα κείμενο, κάποια έκθεση όσον αφορά την ε, εφαρμογή των διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων για ανάπτυξη και ανθρωπιστική δράση, ε, για κάποιο είδους ε, προτάσεις για το μέλλον, ο υποφαινόμενος επίσης έχει αναλάβει μια τέτοια γνωμοδότηση, ήδη αυτή έχει εγκριθεί. Τέλος να πάμε να δούμε τα, τα επόμενα που θα κάνουμε. Επίσης θα πρέπει τον Μάρτιο να ολοκληρωθεί η μάλλον έγινε, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για την αναπτύξη βοήθεια 12 με 16 και από ό,τι γνωρίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί ένα έγγραφο εργασία. Θα παρουσιάσει ε, τα αποτελέσματα εκείνη τη αξιολόγηση. Προβλέπεται αυτό και τι αμέσω επόμενε εβδομάδε. Οπότε θα ήθελα να δω εάν μπορούμε εμεί ήδη να δούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως στοιχείο αυτής της αξιολόγησης ανθρωπιστική βοήθεια, επομένω 12-16. Πολύ σημαντικό. Και παρουσιάστηκε η υπόθεση της σχέσης ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Τελευταία. Και να δούμε τι μάτα πρόοδου μπορούμε σε αυτό το μέτωπο να σημειώσουμε. Τώρα όσον αφορά την ανθρωπιστική συνάντηση ε, κορυφής της παγκόσμια, εγώ έλαβα μέρος στη συνάντηση του Σεντάι όσον αφορά την πρόληψη συγγνώμη, των φιομηνιών ε, και στην Κωνσταντινούπολη ε, που ήταν η άλλη ανθρωπιστική συνάντηση κορυφής και η αίσθηση μου ότι στο Σεντάι ξεκίνησε ένας μηχανισμός αξιολόγησης περιοδικού χαρακτήρα οδήγησε στο Κανκούν δύο χρόνια μετά. Τελικά θα πάμε και στην Γενέβη σύντομα για να δούμε με αυτό το μηχανισμό πώς θα υλοποιηθούν κάποια προγράμματα, κάποιες στρατηγικές. Ό,τι εγκρίθηκε στο Σεντάι για την πρόληψη των κινδύνων. Όμως την ανθρωπιστική κρίση δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, οπότε προχωρούσαμε στα τυφλά. Άρα είναι θέμα τώρα του πώς θα υλοποιήσουμε, πώς θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων θεωρώ ότι είναι θετικό το να έχουμε αξιολόγηση. Και ας μην υπάρχει όπως το για το Σεντάι υποχρεωτικό της, ή μάλλον να είναι υποχρεωτικό το να υποβάλλεται περιοδικά, αλλά θα δούμε πού βρισκόμαστε και έχουμε διάφορους ε, εμπλεκόμενους στην ανθρωπιστική πολιτική που σε σχέση με το Σεντάι ο στόχος είναι να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση πολιτούς χαρακτήρα να υπάρχει πιο πολύ προβλεψιμότητα για την ανθρωπιστική ε, βοήθεια και έτσι αυτή η χρηματοδότηση να δούμε το ότι φρενάρεται φρενάρεται όταν υπάρχει προγραμματισμός εξαμηνίως και μην υπάρχει πολιτής χαρακτήρας όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, αναφέρθηκα στη γνωμοδότηση που κάναμε στην Επιτροπή μας για κάποιο είδους ε, ηρητή υπεράσπιση του ότι τελικά τα ανθρωπιστικά δεν περάσαν στο streamline που έγινε από την Κομισιόν. Ε, και νομίζω συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Άρα είναι σημαντικό να έχει αυτόνομο χαρακτήρα η ανθρωπιστική πολιτική. Επίσης, θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε το μέσο αυτό για άλλους στόχους. Να μην χρησιμοποιείται για άλλα πράγματα πέραν των ανθρωπιστικών και των ανθρωπιστικών κρίσεων. Βεβαίως και θέλουμε να υπάρξει ευελιξία και θεωρούμε θετικό ότι προβλέπεται αύξηση πρικοδότησης 30 με 40% ετησίως. Πρόκειψε αυτό από τις προτάσεις της ε, Κομισιόν. Και άρα στο υπόλοιπο αυτής της θητείας το Κοινοβούλιο για τον επόμενο προϋπολογισμό μη και με τη βοήθεια της Επιτροπής σας θα προβεί σε αυτήν την αύξηση των κονδυλίων για την ανθρωπιστική βοήθεια. Να μην μακρηγορήσω, γιατί και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να λαβούν το λόγο. Αλλά, για να δούμε με λίγα λόγια, τι μπορεί να προκύψει τι μπορεί να γίνει. με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πολλές φορές καλείται να βοηθήσει για κατεπίξεις καταστάσεις και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μια που από ό,τι φαίνεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης πρόκειται να ενταχθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και πάλι ευχαριστούμε για όλη αυτή την πλούσια ενημέρωση για όλες αυτές τις ανθρωπιστικές κρίσεις παντού σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς αυτές οι κρίσεις σοβούν παντού. Τη Δευτέρα σας περιμένουμε στη Μαδρίτη. Και μια υπέροχη τοποθεσία το ώστε αν έχετε την ευκαιρία να περάσετε και το Σαββατοκύριακο. Αλλά εν πάση και αν μείνετε εκεί Σαββατοκύριακο Δευτέρα το πρωί μετά την, ε, μετά την, την, την, την δουλειά, μετά το γεύμα, θα, θα πάμε στο Ρετήρο, ένα ε, υπέροχο ανοιξιάτικο πάρκο της Μαδρίτης και άλλωστε το λέμε αυτό στη χώρα μας ότι το, το Μάρτιο έχει αέρα ε, και τον Απρίλιο έχει βροχές αλλά ο Μάιος είναι υπέροχος Επίτροπε, έχετε ε, την ευκαιρία λοιπόν να πάτε να δείτε το ε, ε, πανέμορφο πάρκο Ρετήρο στη Μαδρίτη. Ποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ε, στη κατάλογο έχω διάφορους. And I have Charles Goins. Does anybody else wish to take the floor? No, I think it's everybody who's here. Ποιος θα ήθελε λοιπόν να πάρει το λόγο. Ξεκινάμε. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, Επιτρόπε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα και που μας μιλήσατε για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στην Ασία, για τα διάφορα προβλήματα, τις ε, δραματικές καταστάσεις στις διάφορες χώρες. Όπως σας είπα, η, ε, μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας είναι η ασφάλεια, η ασφάλεια των δικών μας επαγγελματιών, των δικών μας ανθρώπων. Απ' την άλλη, είναι σημαντικό είναι να ε, τηρείται το διεθνές δίκαιο. Ε, έμαθα τους τελευταίους μήνες για τα διάφορα σκάνδαλα όπου εμπλέκονται επαγγελματίες υγείας και μέλη των ειρηνευτικών αποστολών. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε, αλλά και να προστατεύουμε τους ε, ντόπιου ε, πληθυσμούς. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Η ερώτησή μου είναι η εξής. τι ε, μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να ε, αποφύγει τέτοιες ε, καταστάσεις και τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει σε θύματα τέτοιων καταχρήσεων και κακοποιήσεων. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για την απουσία προγράμματος δράσης, ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την ανθρωπιστική βοήθεια και την κάλυψη των διαφόρων ανησυχιών. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για, την, για τον καθορισμό ενός νέου προγράμματος δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Η Λόρα Σάντσετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πολύ Λίντα και ευχαριστούμε και εσάς κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Έχω μια παρατήρηση και ερώτηση όσον αφορά την συνολική αξιολόγηση για την ανθρωπιστική βοήθεια αυτή που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο. Έχετε πέντε στρατηγικές συστάσεις στην έκθεση όσον αφορά την πολιετή ε, χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα και όσον αφορά την τολμηρή ε, πολιτική και αποτελεσματικότητα. Δεν θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές λόγω των ε, ε, συστάσεων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πώς βλέπετε ε, τον ρόλο των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών πώς θα γίνει η εταιρική σχέση γιατί προβληματιζόμαστε για κάποιες τέτοιες συνεργασίες που έχουν σχέση με ανθρωπιστική βοήθεια πολλές φορέ πρετανεύει η οικονομική ωφέλεια και όχι η ανθρωπιστική ανάγκη. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ότι πλέον δεν θα έχει κάποιες χρηματοοικονομικές ε, ε αρμοδιότητες η DG που τις είχε επί δεκαετίες. Είπαμε ότι δεν έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση, αλλά έχει αυξηθεί, έχει διπλασιαστεί ο αριθμό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Τι θα γίνει με, τη, με τα συμπληρώματα τα δημοσιονομικά, τι θα κάνετε. Πώς θα είναι καλύτερη προοικοδότηση των χρηματοοικονομικών μέσων που χρειάζονται. Just, just to underline the... Θα ήθελα να τονίσω το θέμα τους ε, πολίτους ε, χρηματοδότης από την ΕΚΟ. Ήμασταν στην Ουγκάντα την προηγούμενη εβδομάδα και από ό,τι καταλάβαμε υπάρχει μια ε, κατανομή κονδυλίων σε τήσια βάση σε κάθε χώρα και κατά τη διάρκεια του έτους διατίθενται επιπλέον κονδύλια για να αντιμετωπιστούν εκτακτές καταστάσεις. Κάθε σύμβαση όμως έχει διάρκεια ενός έτους. Πολύ γραφειοκρατία λοιπόν, ε, συνεχής κύκλος γραφειοκρατίας. Και ε, τώρα με, το, με τα νέα προγράμματα έχουμε την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε το σύνδεσμο και να μην έχουμε πια αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά με χρηματοδότηση σε τίσια βάση, ανανέωση κάθε χρόνο. Ε, θα δούμε αλλαγή προκειμένου ε, οι δράσεις μας να είναι πιο αποτελεσματικές. Και τώρα ο Σάρλ έχει το λόγο ένα άτομο από κάθε ομάδα μιλάει και μετά θα μιλήσουμε με τους υπόλοιπους. Ναι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σιλιανίδη για την εξαιρετική παρουσίασή του. Όχι μόνο η, ε, χρειάζεται ολοένα και περισσότερο ανθρωπιστική βοήθεια και αυξάνονται οι ανάγκες σε χρηματοδότηση, αλλά και το γενικό πλαίσιο γίνεται όλο ένα και πιο απειλητικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τον αμερόληπτο χαρακτήρα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να περάσουμε. Εμείς ως Επιτροπή πάντα επιμέναμε σε αυτό το σημείο. Ξέρουμε ότι περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Συνένεση. Και αντί να ε, διαπραγματευτούμε μια νέα συνένεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν απειλείται αυτή η διάσταση. Θα προτιμούσα να μην υπάρχει καθόλου νέα συνένεση, παρά να απειληθούν τα κεκτημένα που ε, ε, κανείς δεν θέλει να αμφισβητήσει στο σημερινό, στη σημερινή συνένεση, στα πλαίσια της σημερινής Μιλήσατε για την επιδημία έμπολα που εμφανίζεται και πάλι στο Κονγκό. Πολύ σημαντικό. Ψηφίσαμε, υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα πριν από μερικά χρόνια. Και φυσικά σε αυτό τονίσαμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες των χωρών που απειλούνται από τον ιό έμπολα, αλλά και ε, τονίζουν το ανθρωπιστικό σύστημα και την αναπτυχιακή πολιτική γενικά. Πολλά έχουμε να πούμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι ουσιαστικά ζητήματα που ήθελα να αναφέρω. Όσο για τα υπόλοιπα, ε, σας στηρίζει η Κομισιόν, καθώς και η πολιτική μου ομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει εξαιρετική δουλειά στο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, ίσως θα ήταν καλό να ε, απαντήσει ο Επίτροπος και μετά να ακουστούν και οι επόμενες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ε, ε παρατηρήσεις, τα σχόλια του φίλου μου, κ. Σαλόν. Σας ευχαριστώ πολύ για ε, την έκθεσή σας. Είμαι πεπισμένος ότι οι παρατηρήσεις σας θέτουν ε, στη καρδιά των συζητήσεων πολλά από τα κοινά μας προβλήματα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως σας είπα. Χαίρομαι που η πρόταση για το νέο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνει μια σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την ανθρωπιστική βοήθεια. Προτείνουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για την επόμενη 7 1,5 δισεκατομμύρια 11,5 ευρώ, 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε όλη την 7 ε, 1,5 ε, εκατομμύρια κάθε χρόνο. Πολύ σημαντική αύξηση ε, αυτή της ενής, των κονδυλίων για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά υπάρχουν και επιπλέον ε, στοιχεία που ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Είναι σημαντική η ευελιξία, το είπατε. Γι' αυτό λοιπόν ο μηχανισμός έκτακτης βοήθειας θα παραμένει διαθέσιμο και το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για εξωτερική δράση θα χρηματοδοτήσει το σύνδεσμο. Προβλέπετε λοιπόν επιπλέον ευελιξία για τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρόκειται για κάτι καινούριο στα πλαίσια των προσπαθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, ε, καταστάσεις χωρίς προηγούμενο, όπως είπατε. επιμείνατε στο παγκο... στην παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και στη Σεντάι και στο Κανκούν. Προτείνατε ήδη κάποιο μηχανισμό για την αξιολόγηση της υλοποίησης των ε, προτάσεων και του πλαισίου. Καλή ιδέα, σίγουρα. Πρέπει να δούμε πώς ε, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Χρειαζόμαστε ένα ε, σύστημα ελέγχου, αλλά όπως ε, συζητήσαμε πολλές φορές με τους συνομιλητές μου και ε, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, κάποιες φορές υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο πλαίσιο που έχει ε, συμφωνηθεί για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την ε, πολιτική προστασία από τη μία και από την άλλη την εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Νομίζω ότι είναι καλό να συζητώνται αυτές οι προτάσεις ε, σχετικά με την αξιολόγηση στα πλαίσια του συστήματος του ΟΗΕ προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία για να δούμε μαζί πώς μπορούμε να ε, επισπεύσουμε την εφαρμογή αυτής της ιδέας. Η πρότασή σας ε, για κάποιες ευχάριστες δραστηριότητες και χαλάρωση στη Μαδρίτη είναι ευπρόσδεκτες, αλλά γνωρίζετε ότι δεν θα έχω ε, χρόνο για τέτοιες δραστηριότητες, ε, γιατί θα φτάσω στη Μαδρίτη αργά την Κυριακή. Ρωτήσατε για την έκθεση της αξιολόγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας για το διάστημα 2012-2016. Αυτή η έκθεση έχει ήδη δημοσιευτεί τονίζει ότι η ανθρωπιστική ε, βοήθεια που προσφέρεται είναι κατάλληλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δράση της προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία. Το διαπιστώσαμε χάρη στις δραστηριότητές μας ε, επιτόπου. Και θα ήθελα επίσης να σας ε, συγχαρώ για την εξαιρετική έκθεσή σας. Φυσικά υπάρχουν ε, πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Πιστεύω πάντως ότι αυτή η έκθεση αξιολόγησης που έχει δημοσιευτεί θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των δικών μας δράσεων στον ανθρωπιστικό τομέα. Αγαπητοί φίλοι, επιμείνατε στη σημασία της πρόληψης και ε, της τήρησης ε, της ε, εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, ανθρωπιστικού δικαίου επιτόπου. Σίγουρα κάποιοι από εσά έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από μένα επιτόπου. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Κατά τη διάρκεια των διαφόρων ταξιδιών μου, επισκέψεών μου, διαπίστωσα επιτόπου ότι δυστυχώς σε πολλές περιοχές που πλήττονται από κρίσεις επικρατεί απόλυτη ε, ανασφάλεια ε, όχι μόνο για τους επαγγελματίες υγείας και τους, ε, τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά για όλα τα άτομα που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Διάφορες οργανώσεις όπως ε, η Oxfam, άτομα που εργάζονται για αυτές τις ε, οργανώσεις ε, έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα τα οποία οποία πειράζουν αρνητικά την ε, δική μας εικόνα. Προσωπικά είμαι κατηγορηματικός. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή σε περίπτωση ε, ε, υποψίας λανθασμένων χειρισμών, τέτοιων, τέτοιων χειρισμών από μέλη ε, συνεργαζόμενων οργανώσεων, όλοι οι εταίροι πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα. Οι ε, συμβάσεις που υπογράφουμε προβλέπουν ε, δεσμευτικές, ε, δεσμευτικούς όρους μετά από του, ε, τους ισχυρισμούς που γνωστοποιήθηκαν το Φεβρουάριο για σεξουαλική κακοποίηση ζητήσαμε από τους εταίρους μας να μας δώσουν ε, στοιχεία για το πώς αντιμετωπίζουν, πώς προλαμβάνουν ε, τέτοιες συμπεριφορές. Περιμένουμε ε, ακόμα κάποιες ε, ε, απαντήσεις. Στο μεταξύ, οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ εξετάζουν τις απαντήσεις που έχουν λάβει ήδη και φυσικά συντονίζουμε τις δράσεις μας και με άλλους δωρητές. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Συζητήσαμε αυτό το θέμα. Συζήτησα και με τον Φίλιππο Γκάντι, με τον Πιλιουνάνε στην Γενέβη και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει ε, να ανακτήσει η ανθρωπιστική ε, κοινότητα την ε, θετική της εικόνα. Γιατί αυτά τα λίγα περιστατικά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και στα πλαίσια της επικοινωνίας μας με τους πολίτες. Συνένεση και πρόγραμμα δράσης. Η συνένεση, η Ευρωπαϊκή Συνένεση είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρωπιστική μας δράση. Είμαστε πεπισμένοι ότι η τήρηση αυτών των αρχών είναι ε, πρωταρχική σημασία για τις δράσεις μας στο στην παγκόσμια ε, διάσκεψη, ανθρωπιστική διάσκεψη ε, υπήρξε συνένεση σχετικά με τη σημασία αυτής της, ε, της στήριξης αυτών των αρχών. Είμαι υπέρ της δράσης, όχι λόγια. Πρέπει να μετατρέψουμε τα λόγια σε δράσεις επιτόπου. Και αυτό που είναι πιο, ακόμα πιο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε ότι ε, υπάρχει συνένεση ε, για την ανθρωπιστική ε, δράση και ότι τηράνται κάποιες αρχές επιτόπου. Είναι καλύτερο αυτό από το να υπάρξουν επιπλέον γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που αυξάνουν την γραφειοκρατία και δεν προσφέρουν καμία προστιθέμενη αξία. Ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να αποφύγουμε την δημιουργία νέων γραφειοκρατικών εμποδίων γιατί αυτό θα μας ε, θα δυσχεραίνει το έργο μας στην πράξη. Έμπολα. My Όσο για τον έμπολα. Ο αγαπητός φίλος κύριος Γκέριντς ε, και εγώ συνεργαζόμαστε για να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης στην περασμένη φορά που είχαμε κρούσματα στη Λιβερία, τη Γουινέα και τη Σιέρα Λεόνα. Και γνωρίζετε ότι χάρη στην δική σας έκθεση είδαμε πως ε, δυστυχώς ήμασταν εκτός πραγματικότητας και αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα την εποχή εκείνη. Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα. Όπως σας είπα, είμαι σε συνεχή επαφή με τον ε, ομόλογο μου για τα θέματα αυτά. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε δύσβατες περιοχές. Υπάρχουν 42 κρούσματα μέχρι τώρα, τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα μόνο, 20 πιθανά κρούσματα έμπολα και 19 με υποψία έμπολα. Έχουν σημειωθεί θάνατοι. Χθες 15 Μαΐου δεν είχαμε κάποια νέα ειδοποίηση για νεοκρούσματα. κρούσματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα τρία υποψήφια εμβόλια. Έχει διαθέσει γι' αυτό ένα αρκετά σημαντικό ποσό, αλλά και πάλι το ύψος της βοήθειας ε, θεωρείται αρκετά χαμηλό. Με τον Γενικό Διευθυντή κύριο Ντέδρος, είμαστε συνέχεια σε επαφή για να δούμε αν μπορέσουμε να διαθέσουμε μερικά κονδύλια από τη δική μας χρηματοδότηση για να διατηρήσουμε αυτή την αερογέφυρα ανάμεσα στην Κινσάσα και στις περιοχές αυτές που έχουν σημειωθεί τα κρούσματα. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η νέα χρηματοδότησή μας και όπως είπα, ακριβώς εξαιτίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Ιατρών την περασμένη φορά που σημειώθηκαν κρούσματα πριν από τρία χρόνια. Αυτή τη φορά είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι έτσι ώστε να μπορούμε να παράσχουμε βοήθεια και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες επιτόπου και να έχουμε καλύτερη ε, δυνατότητα πρόβλεψης της κατάστασης. Νομίζω πως λίγο πολύ ήδη απάντησα στις ερωτήσεις σας, ε, αγαπητοί συνάδελφε, για, την, το σύνδεσμο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και επίτρεψέ μου Λίντα να πω για την Ουγκάντα ότι γνωρίζεις τη δυσκολία της ε, συνέχισης της χρηματοδότησης. Μόνο 5-6% των ε, προγραμμάτων συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται πάνω από ένα έτος. Γνωρίζω πως σε απασχολεί πολύ αυτό το θέμα και θέλω να πω ότι και εγώ με το επιτελείο μου συζητάμε ε, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα επιτόπου ακριβώς γιατί οι καταπήγουσες ανάγκες είναι δύσκολο να ε, προβλεφθούν. Και είναι ακριβώς ε, αυτή η δυσκολία για, στη χρηματοδότηση. Είναι πολύ δύσκολο να ε, εγκριθεί χρηματοδότηση βασισμένη σε προβλέψεις των αναγκών που θα προκύψουν. Γιατί τα προγράμματά μας δεν ασχολούνται μόνο με το να προβλέπουν τις ε, πιθανές μελλοντικές ανάγκες, αλλά και ε, με τις ε, υφιστάμενες και γι' αυτό υπάρχει δυσκολία να εγκριθεί χρηματοδότηση για πάνω από ένα χρόνο, να συνεχιστεί ένα πρόγραμμα πάνω από ένα χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χιμένα θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Στα Ισπανικά. Στη μητρική μου σας τα από τα Ισπανικά. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας και συντονιστείτε στο κανάλι 8. Σας ευχαριστώ για το έργο σας. Δεν έχουμε καμία εμφιβολή ότι ε, ασχολείστε με μεγάλη ζέση. Επίσης σας ευχαριστώ για αυτή την αύξηση του 30%. Αυτή την αύξηση που προκεινοφελίζει πάρα πολύ κόσμο και θα ήθελα να σας πω ότι 100% συμφωνώ με όλα όσα έχετε πει για τον ε, Λίβανο. Ε, για το ότι ο Λίβανος ε, φυσικά έχει υποδεχθεί τους μισούς πρόσφυγες και ξέρετε μόλις επέστρεψα από την Κύπρο την πατρίδα σας την αγαπώ πάρα πολύ και όσον αφορά το Κυπριακό πάντοτε μιλούμε όσον αφορά τους πρόσφυγες αλλά μιλούμε εκεί για πρόσφυγες Ευρωπαίους. Πήγαμε στην παραλία, στην Αμόχωστο και εκεί ε, είδαμε για κάποιους που είναι πρόσφυγες 44 χρόνια, είναι με, το, με τη βαλίτσα στο χέρι και δεν έχουν ε, ζητήσει. Δηλαδή φύγανε ενώ ο λόγος είχα, ετοίμαζαν ε, καφέ ξαφνικά. Τους στηρίξαμε, τους, τους, τους συζητήσαμε και επίσης κάτι που αναφέρεται είναι σημαντικό. Μας αναφέρεται την ανθρωπιστική κρίση στην Βενεζουέλα. Βοηθούμε την Κολομβία, βοηθούμε την Βενεζουέλα. Θέλετε να μου πείτε πιο συγκεκριμένα δύο λόγια. Τι γίνεται με το Μαδούρο. Τι γίνεται με τη βοήθεια. Έχω πάει εκεί και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει κανένα ότι έφτασε σε, σε, σε τόση δυστυχία μια τόσο πλούσια χώρα γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα για τα παιδιά. Οπότε, εάν μπορείτε, πέστε μας, υπάρχει τρόπος να τα καταφέρετε. Επίσης, όσον αφορά την Νιγηρία. Ξέρουμε ότι επέστρεψαν ε, τα κορίτσια που είχε απαγάγει η Μπόκο Χαράμ. Τι γίνεται τρόμος με το μέτωπο ασφάλεια εκεί. Ε, μια που εκεί πέρα ε, θεωρούν και αυτό, αυτό λέει η Μπόκο Χαράμ ότι όποιος δεν είναι Ισλαμιστής και, κάνει αμαρτία. Τώρα επίσης για το τελευταίο που μας ε, αναφέρατε ε, για την Σιέρα Λεόνε. Τι γίνεται με την εκπόρνευση των κοριτσιών και τι γίνεται και με αυτό το βίντεο που είδαμε από τους καλόγερους. Ζουν στο δρόμο αυτά τα κορίτσια που εκπορνεύονται και υποφέρουν. Και πάνε σε κάποια ε, πλωτά μπαρ για να εξυπηρετήσουν σε εισαγωγικά τους Κινέζους εργαζόμενους εκεί. Θα πρέπει κάτι να συνοήσουμε τις εκεί αρχές για να σταματήσει αυτή η κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας συναντήσω θα είμαι στην ε, Μαδρίτη να πάτε κι εσείς. Δεν ξέρω θα, δεν θα μπορέσω να σας πάω βόλτα να σας συνοδεύσω στο ρετήρο όπως είπε ο, ο φίλος ε, Ενρίκε. Δεν πειράζει, θα δούμε. Και ίσως ε, να μπορέσουμε να κάνουμε τη βολτίτσα αν τελικά σας περισσέψει λίγος χρόνος. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η Αλισλάιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ε, ολοκληρωμένη εικόνα που μας δώσατε, για αυτά που έχουν γίνει και για αυτά που πρέπει να γίνουν. Τρία πράγματα θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, είναι σαφές ότι δεδομένων των νέων πολιτικών συνθήκων η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να ηγηθούμε και στην αναπτυξιακή βοήθεια και στην ανθρωπιστική βοήθεια, διότι χωρίς εμάς κανείς άλλος δεν πρόκειται να αναλάβει δράση. Έπειτα, άκουσα τον ε, κύριο Γκέρεν το πρωί ο οποίος ήταν αγανακτισμένος για την ε, έλλειψη υλοποίησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν πολλές χώρες σε διεθνές επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Μετά, δεύτερον, η ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Ε, αναφερθήκατε ε, στην περίπτωση της Ελλάδας, την οποία φυσικά και στηρίξαμε, όμως πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, ιδιαίτερα ε, στην περίπτωση της οδού της Μεσογείου και δεν θα σταματήσω να επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση στις περιπτώσεις διάσωσης, ειδικά διάσωσης στη θάλασσα τα προγράμματα Σοφία και Τρίτον σώζουν ζωές. Χρειάζεται όμως πλήρη σε ανθρωπιστική εντολή έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή. Τρίτον, όπως είπε και η Λίντα, στην ε, περίπτωση της Ουγκάντα πρέπει να γίνει περισσότερα. Έχουμε 1,4 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ουγκάντα. Η Ουγκάντα έχει μία αρκετά προοδευτική πολιτική, την οποία νομίζω πως γνωρίζετε, γιατί έχετε βρεθεί εκεί. Η πολιτική της είναι ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές και οι πρόσφυγες που φτάνουν παίρνουν ένα κομμάτι γης για να ε, εγκατασταθούν. Δείχνει αλληλεγγύη η Ουγγάντα και μάλιστα ένας ε, τοπικός ηγέτης σε, μια, ένα καταβλισμό στο βόρειο τμήμα της Ουγγάντας μας είπε ότι καλωσορίζουμε τους πρόσφυγες και αποφασίσαμε να μοιραστούμε τη γη μας μαζί τους και να δουλέψουμε μαζί έτσι ώστε μια μέρα να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους όχι ως ζητιάνοι αλλά με αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Παράλληλα επισκεφθήκαμε διάφορα έργα και προγράμματα τα οποία έχουν στόχο να προωθήσουν την κοινωνική συνοχή τόσο των ε, κοινοτήτων προσφύγων όσο και των ε, τοπικών κοινοτήτων στις οποίες ε, βρίσκονται. Είναι τεράστια η προσπάθεια που καταβάλλεται για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Είναι προγράμματα που αλλάζουν ζωές, όμως ε, η ανθρωπιστική κρίση πάσχει από υποχρηματοδότηση. Μόνο το 6% των προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτείται. Και αν λάβουμε μάλιστα υπόψη την ε, αστάθεια στην περιοχή, στο Κονγκό, στο Μπουρούντι που τα πράγματα είναι ανησυχητικά, στο Νότιο Σουδάν που είναι τραγική η κατάσταση δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε αυτήν την ε, προοδευτική πολιτική, να τη στηρίξουμε την πολιτική της Ουγκάντα ιδιαίτερα σε θέματα υγείας, σε θέματα επιστημιστικά, διότι γνωρίζετε πως υπάρχουν τρομερές δυσκολίες ε, για τη σύντηση των ε, προσφύγων. Πρέπει τον Ιούνιο να μειώσουν τις μερίδες φαγητού και αυτό θα είναι καταστροφικό μετά εκπαίδευση, παιδεία είναι και εκεί προβληματική κατάσταση. Το 86% όλων των προσφύγων είναι γυναικόπαιδα και πρέπει να φροντίσουμε για ε, την μόρφωσή τους. Και έπειτα, όπως είπε και η Λίντα, θα πρέπει να αναλογιστούμε αν χρειαζόμαστε πολιετή χρηματοδότηση και κατά πόσο, διότι βλέπουμε ότι στην περίπτωση της Ουγκάντα χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμός και σιγουριά. Και σίγουρα η χρηματοδότησή μας πρέπει να είναι σε θέση να διατίθεται μακροπρόθεσμα. Αυτά από μένα προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, θα υπάρξει μια αποστολή. Νομίζω και εσείς θα πάτε. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε την παρουσία μας εκεί, έτσι ώστε να δείξουμε και στην κυβέρνηση ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που θα πάτε εκεί. Και όπως είπατε, η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για τους πρόσφυγες στην Ουγκάντα, ιδιαίτερα όμως η ποιοτική εκπαίδευση. Έχουμε διαπιστώσει πόσο δύσκολο είναι αυτό στην πράξη, διότι ξέρετε πολλές φορές ε, είναι ένα κουτάκι που πρέπει να συμπληρώσουμε, ότι ναι ε, γίνονται μαθήματα στα παιδιά. Όμως η πραγματικότητα πολλές φορές απέχει κατά πολύ από ε, αυτό το κουτάκι που συμπληρώνουμε. Γιατί μιλάμε με τους δασκάλους και μας λένε ότι οι τάξεις αποτελούνται πολλές φορές από 100-150 παιδιά. Είναι αδύνατον σχεδόν να παρασκευθεί επαρκή εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλές γυναίκες πρόσφυγες που θέλουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, δεν έχουν όμως ε, χρήματα, δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν μπορούν να πληρώσουν για τα παιδιά τους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ε, προβλήματα και πολλές ελλείψεις στην εκπαίδευση και πρέπει σίγουρα να το έχουμε αυτό κατά νου και να μην χάνουμε το στόχο. Υπάρχουν κάποια προγράμματα για νέους, κατάρτισης, για παράδειγμα κατάρτιση μηχανικού αυτοκινήτων για τους νέους και στην Ουγκάντα και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το προσωπικό της ε, ΓΔ ΕΚΟ έχει κάνει τρομερή δουλειά. Στη Βόρεια Ουγγάντα μένουν σε σκηνές οι πρόσφυγες, σε άθλιες συνθήκες. Ζητάμε από τους γιατρούς να εγκαταλείψουν τα πάντα και να πάνε εκεί, αλλά πρέπει να, του να τους προσέξουμε, διότι όταν κάποιος ε, θυσιάζει την προσωπική του ζωή για να πάει εκεί, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί. Οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι καλές. Και γνωρίζουμε επίσης πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα PIS. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε για την ε, διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Τώρα, ε, ξέρω πως ε, για το εμβόλιο κατά το εμπόλα ε, αρμόδιος είναι ο Επίτροπος Αντριουκάητη, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε εσεί κάτι γι' αυτό. Και τέλος, οι συνολικές δαπάνε για την διάθεση χρηματοδότησης προσυλλοποίηση των στόχων της Αντίσα Μπέμπα, ούτε στο ελάχιστο δεν φτάνει αυτή που χρειάζεται ιδιαίτερα στην περίπτωση των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών, διότι έχει δοθεί έμφαση στην ε, Μέση Ανατολή και ο στόχος του 0,2% δεν μπορεί να επιτευχθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν την Αφρική και την κρίση εκεί, ακόμα και αν αυξάνονται οι απαιτήσει. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη, νομίζω πως ναι, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ερωτήσεις μου έστειλε επιστολή το Συμβούλιο Προσφύγων της Νορβηγίας και ήταν πολύ ενισχυτικά αυτά που διάβασα. Μου είπε ότι καταστρέφεται το πρόγραμμα, καταργεί τη χρηματοδότηση. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Μετά, να παραδεχτούμε βέβαια ότι κάθε φορά πηγαίνουμε αποστολή σε ένα μέρο γυρίζουμε και λέμε ότι αυτό είναι χώρα προτεραιότητας και θέλουμε να δώσουμε προσοχή. Όμως θα σταματήσω εδώ και θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε σε αυτά στις τελικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Δίχως αμφιβολία συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες σας και έχω τις ίδιες προτεραιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο την εκπαίδευση. Δεν είναι απαραίτητη μόνο η εκπαίδευση ως όχημα πολιτικής προστασίας, αλλά η σημασία έχει η εκπαίδευση να είναι ποιοτική. Διότι πρέπει να είναι το όχημα που θα βοηθήσει τα παιδιά να πάνε πέρα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, να σπουδάσουν. Και επομένω, με τη δική σας στήριξη καταφέραμε να αυξήσουμε κατά 8 φορές τον προϋπολογισμό μας. Και προτού λήξει η θητεία μου, οφείλω να ομολογήσω ότι θα ήθελα να αυξηθεί λίγο περισσότερη χρηματοδότηση. Είναι βέβαια κάτι που εξαρτάται από την ε, διαθεσιμότητα των κονδυλίων, όμως έχω δει από την πείρα μου πως ε, από τα πολλά προβλήματα και από τα πολλά ζητήματα η έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες όλων των ε, εξαναγκαστικών των ε, καταναγκαστικών γάμων, της ε, ριζοσπαστικοποίησης, στρατολόγηση, τρομοκρατία. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να συνδεθεί η εκπαίδευση με τα εθνικά προγράμματα. Ουγκάντα τώρα. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι υποδειγματική η περίπτωση της Ουγκάντα στην υποδοχή των προσφύγων, ακριβώς γιατί, όπως είπατε και εσείς, δίνουν γη στους πρόσφυγες. Τώρα, στην Ευρώπη, ας αναρωτηθούμε αν είναι εύκολο να ακολουθήσουμε το ίδιο μοντέλο με την Ουγκάντα. Ε, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, ο χώρος που έχουμε είναι τόσο περιορισμένος που δεν γίνεται αυτό. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι κάθε χώρα μπορεί να ακολουθήσει το δικό της προσαρμοσμένο μοντέλο και αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Πρέπει να βρούμε τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην ανθρωπιστική βοήθεια και πώς μπορεί αυτή να δοθεί δεδομένων των ε, ιδιαιτερότητων αυτών της κάθε χώρας. Βέβαια. Όταν πήγα ο ίδιος στην Ουγκάντα, είδα με τα μάτια μου αυτήν την εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στις κοινότητες που φιλοξενούν πρόσφυγες και τους ίδιους τους πρόσφυγες. Γι' αυτό δώσαμε έμφαση σε αυτό και μέσω διαφόρων προγραμμάτων σίγουρα αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι η καλύτερη δυνατή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τις τοπικές οικονομίες και να δείξουμε στις τοπικές ε, κοινότητες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους σκέφτεται, δεν τους έχει εγκαταλείψει. Πήγα και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, μέσα στην Ευρώπη και τα είδα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Και ακριβώ επειδή επισημάνατε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνη της στην αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κατάστασης, να σας ε, ομολογήσω ότι πολλές φορές αισθανόμαστε μόνοι ως Ευρωπαίοι και είναι αρκετά οδυνηρή η εμπειρία στην ε, σύνοδο για την στην Ουγγάντα, νομίζω πέρυσι τον Ιούνιο, όταν υποσχεθήκαμε να διαθέσουμε 85 εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη και η... τα κονδύλια που διατέθηκαν ήταν το 82% του συνόλου της βοήθειας που υποσχέθηκαν όλα τα κράτη στη γη. Πού είναι λοιπόν όλοι αυτοί. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν αισθάνομαι υπερήφανος για τους πολίτες μας, διότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ανθρωπιστική βοήθεια στηρίζεται μέσω της συνένεσης και οι πολίτες αισθάνονται υπερήφανοι για τη συνεισφορά τους αυτή για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Βενεζουέλα τώρα. και Κολομβία. Φυσικά και συμμερίζομαι την... τα συναισθήματά σας ε, και στην περίπτωση των συμβάντων στη Σιέρα Λεόνε. Δυστυχώς είναι αναπόφευκτο να παρατηρούμε τέτοια περιστατικά σε πολλές περιοχές που μαστίζονται από κρίσεις, από ένδια κτλ. Ο στόχος μας γενικότερα είναι να βρούμε ανθρω... εταίρους ανθρωπιστικής βοήθειας επί τόπου, πρώτον για να αποτρέψουμε ε, την εμφάνιση νέων κρίσεων μέσω της εκπαίδευσης και με άλλους τρόπους, αλλά και με την συνεχόμενη παροχή στήριξη στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Όταν πήγα στη Κολομβία και τη Βενεζουέλα, Ανακοινώθηκε, όπως είπατε και εσείς, ε, πρόσθετη χρηματοδότηση. Συναντηθήκαμε λοιπόν με τους εταίρους μας και συμφωνήσαμε για την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων στη Βελεζουέλα ανεξάρτητα με το αν, αρνήθηκε η κυβέρνηση να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Νομίζω πως υπάρχει μια σιωπηλή συνένεση και ήδη έχουν αποδεχτεί πολλές ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα ε, στη... στον ιατρικό τομέα και στην ε, παροχή φαρμάκων. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις εκεί Πιστεύω όμως ακράδαντα και αυτό επιτρέψτε μου να το θεωρήσω πολιτική άποψη πως η πιο σημαντική εξέλιξη είναι αυτά τα εξαιρετικά προγράμματα για εθνική συμφιλίωση με την ε, ηγεσία του Σάντος διότι η Κολομβία είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Είναι η πιο σημαντική χώρα. Και μέσω της ε, διαδικασίας συμφιλίωσης και της σταθεροποίησης της Κολομβίας θα δούμε αυτό να έχει θετικές επιπτώσεις και σε όλη την περιοχή. Επιτρέψτε μου τώρα να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα, διότι θα ήθελα να χρησιμοποιήσω λεξιλόγιο και ορολογία ιατρική. Λίντα, ε, το θέμα του βαξίν φορέμπολα. Γνωρίζετε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια επικεντρωθήκαμε στη δημιουργία του εμβολίου. Ε, δώσαμε όντως πολλά λεφτά για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Ε, προσωπικά θεωρώ και από τις ιατρικές μου γνώσεις ότι ε, το εμβόλιο είναι Όντω αποτελεσματικό, όπως χρειάζεται χρόνο και να αποδειχθεί με βάση τα medical standards. Ε, και ο, ο φίλος και συνάδελφος ο Τέτρος από το WHO ε, με ενημέρωσε εχθές ότι έχουν ήδη αρχίσει να παρέχουν το εμβόλιο όχι μόνο σε humanitarian workers αλλά και σε πληθυσμούς στην περιοχή που τώρα είναι ε, επηρεασμένοι από τα πρώτα κρούσματα έμπολα. Ε, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό test case που θα δούμε τα αποτελέσματα on the ground αλλά ε, θα επιμείνω σε αυτό που είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση. Είμαστε ως παγκόσμια κοινότητα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλύτερα προετοιμασμένη σήμερα παρά τρία χρόνια πριν. In all angles of the Ebola και επειδή δημιουργήσαμε το EU Ebola EU Medical Corps ε, είμαστε έτοιμοι και στο ΜΕΤΕΒΑΚ και σε όλες τις ε, περιπτώσεις να αντιδράσουμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και να αποτρέψουμε επέκταση της επιδημίας. Ε, όμως πρέπει να είμαστε alert, no complacency on Ebola ε, και γι' αυτό είμαστε σε συνεχή επαφή με τον ε, WHO για να αποφύγουμε οτιδήποτε πιο δυσάρεστο. Thank you so much uh, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, πολύ ευχάριστη ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα ε, που μοιράστηκα μαζί σας αυτές τις εξαιρετικές παρατηρήσεις ε, και τα σχόλια. Πρέπει να βελτιώσουμε τους την, αυτού μας και το ε, σύνολο της δράσης μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Θα ήθελα ε, να σας ευχαριστήσω επίσης και επειδή όταν ήμασταν στην Ουγγάντα μας ε, φιλοξένησε η ΕΚΟ, μας υποδέχτηκε με εξαιρετικό τρόπο και φρόντισε και για τα πρακτικά ζητήματα και τη μεταφορά μας. Συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα και πάμε στο 13. Πολύ θρυβερό για μένα γιατί πρώτα μιλήσουμε για την αναπτυξιακή βοήθεια Ηνωμένου Βασιλείου Ένωση μετά το Brexit. Τα συζητήσαμε πριν από καιρό αυτά στην Επιτροπή, τότε όμω δεν ήταν το τοπίο πολύ ξεκάθαρο για το τι θα γίνει μετά το Brexit. Ούτε τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν ξεκαθαριστεί. Τι να σας πω για τις διαπραγματεύσεις και πού βρισκόμαστε τα πράγματα. Μα ούτε το τοπίο, το, έσω, το εσωτερικό τέλο πάντων δεν έχει ξεκαθαριστεί στη Βρετανία πάντως. Έχουμε τώρα τα οικονομικά θέματα τα οποία έχουν λυθεί. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τις υποχρεώσεις προς το EDF και σχέση με το ε, πλαίσιο και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής γιατί η κυβέρνηση είπε ότι θέλει να γίνουν όλες οι ρυθμίσεις με ανοιχτό πνεύμα και ε, λέει η κυβέρνηση της Βρετανίας ότι θα πρέπει οι εταίροι μας να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε στατικό επίπεδο κλπ. κλπ. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί ακόμα υπάρχουν διαπραγματεύσεις ένωσης ε, κυβέρνησης. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το non-paper, να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, όπου πάμε ε, στον κόσμο διαπιστώνουμε ότι είναι πρωταγωνιστής της ε, ανάπτυξης προσπάθειας η Αγγλία και έχουμε το 0,7% που συζητήσαμε τι κάνει κάθε χώρα σε σχέση με τις υποχρεώσεις και ήταν πρωταθλήτρια για το 0,7% το Ηνωμένο Βασίλειο παρά τα οικονομικά προβλήματα οπότε θα είναι απώλεια να μην συμμετέχει ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια θα χάσει και η Ευρώπη, θα χάσουν και η Βρετανία. Τώρα, έχουμε καλέσει τον James Μακάι, που είναι επικεφαλής ε, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη διαχείριση της πολιτικής ανάπτυξης και επίσης την Κλέρ Godfrey που ασχολείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με το δίκτυο των ΜΚΟ για την ανάπτυξη. Οπότε θα μας πούν από πλευράς Αγγλίας και από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης τι ισχύει για τις πολιτικές ανάπτυξης. Πρώτος ο Τζέιμς Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και επίσης ευχαριστούμε που μας δώσατε το λόγο εγώ εργάζομαι στο Μάστριτ για το ECDPM, αλλά συμμετέχω και σε κάποια think tanks για την ανάπτυξη. Το ODI στο Λονδίνο, ε, στην, ε, το γερμανικό στη Βόνη, το Ιντρί, στην ε, ε, Γαλλία και κάποιον άλλον ψηφιακό στην Ρώμη. Και όπως είπε η Λίντα Μακάβαν, είναι δύσκολο να συγκεκριμενοποιήσουμε τα πράγματα. Και θα προσπαθήσω τέλος πάντων να σας ενημερώσω, να δούμε κάποια βασικά πέντε σημεία και μετά δούμε ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες για τις διαπραγματεύσεις. Και εσείς όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε στην Ευρωπαϊκή Τροπή. Τώρα, αυτοί οι πέντε βασικοί άξονες χρηματοδότηση, εμπειρογνωμοσύνη, πολιτική επιρροή, κατάτμιση της βοήθειας και ε, οπότε πρώτα πρώτα όσον αφορά την χρηματοδότηση τα πόσα είναι γνωστά θα έχουμε 15% τρίβα στον προπολογισμό 1,5 δις όσον αφορά ε, τον προπολογισμό για την βοήθεια ετησίως ε, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με το σύνολο του ODA της αντισιακής βοήθειας η ανάλυση λέει ότι το 0,7% συνεχίσει να το πληρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο σαφώς, άρα είναι θέμα του πού θα πάνε αυτά τα χρήματα και από πλευράς Ένωσης θα επηρεαστεί η θέση της για την παγκόσμια ψυχική βοήθεια πάει στο 15% και ίσω λίγο πιο κάτω και επίσης η ε, ο στόχος για την αναψυχιακή βοήθεια. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα δύο αρνητικά. Θα πρέπει αυτά να απασχολήσουν την Ένωση. Και βραχυπρόθεσμα, όπως είπε ο Πρόεδρος, θα υπάρξουν λίγες επιπτώσεις, μικρές, περιορισμένες, γιατί θα συνεχίσει να τιμά τις υποχρεώσεις της η Αγγλία όσον αφορά το EDF. Τώρα, να δούμε εάν θέλει αύξηση στον ODA, στο MFM η Ένωση, τότε θα έχουμε συνολικά αύξηση στο ODA. Ανάλογα με το αν θα χρησιμοποιήσουν νέους πόρους τα κράτη-μέλη ή αν θα ρίξουν λεφτά στη, στην Ένωση για τα κόψουν από τις διμερείς προσπάθειες. Οπότε το παγκόσμιο ODA μπορεί να αλλάξει Τώρα για την πολιτική μας, πάντοτε είχε κάποιες προτεραιότητες, η Ένωση και η Αγγλία επίσης. Ε, LDC, φτώχεια, συγκρούσεις, βάλλοντες ε, καταστάσεις και άλλες προτεραιότητες. Αλλά δεν είναι μόνο η Αγγλία πέρα αυτών των προτεραιοτήτων. Και επίσης, πιο μακροπρόθεσμα η απουσία του Ηνωμένου Βασιλείου θα επηρεάσει αυτέ τι προτεραιότητε, θα υπάρξουν αλλαγέ. Οπότε και τα κρατημέρια που θέλουν ίδιε προτεραιότητες θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να παραμείνουν αυτέ οι προτεραιότητες. πάντω. αυτά θα γίνουν ε, από το βράδυ στο πρωί, θα γίνουν πιο μακροπρόθεσμα, αλλά θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Κάτι άλλο είναι το τι γίνεται με τι προτεραιότητε των ΜΕΝ και των ΔΕ. Υπάρχει το ίδιο μήκο κύματο αλλά είπαμε ότι και αυτό θα αλλάξει μακροπρόθεσμα, οπότε η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα δυσκολέψει. Και με αυτή την έννοια μετά το Brexit είναι σημαντικό να κινηθούμε ταχύως για να υπάρχει καλό επίπεδο συνεργασίας. Εμπειρογνωμοσύνη, γνώση, δαπανούνται πάρα πολλά για έρευνα και κλπ. Επομένως ε, όλη αυτή η βρετανική έρευνα δεν θα υπάρχει πια, δεν υπάρχει αυτή η συμβολή στην ευρωπαϊκή συνολική προσπάθεια. Να δούμε αν θα συνεχίσει να θέλει το Μένο Βασίλειο να μεταδώσει τις γνώσεις που αποκτά, άρα εδώ θα υπάρχει κάτι αρνητικό, άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερη προσπάθεια όσον αφορά την ε, έρευνα για τη διαμορφώση των πολιτικών. Πολιτική επιρροή, αυτό σχέση με την παγκόσμια σκηνή, θα υπάρξει απώλεια και από τις δύο πλευρές όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση. Νομίζω αυτό είναι και σαφές για όλους. Και επίσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό πόσο στενή συνεργασία θα έχουν οι δύο πλευρές αν θέλουν να συνεχίσουν να έχουν το ίδιο επίπεδο επιρροή στο πολιτικό γίγνεσθε στο παγκόσμιο σκηνή. Και το τελευταίο σημείο που είναι η εγκατάτμιση της βοήθειας. Σας το λέω αυτό γιατί δεν έχει συζητηθεί. Ε, δεν αναφέρει τόσο πολύ στα έγγραφα που ασχολούν με το Brexit. Θεσμικά όργανα και το ODA αυτών είναι ένας διάβλος για να το προωθήσουν και Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα δημορφωθεί η παγκόσμια συνεργασία γιατί με την βοήθεια αυτήν υπάρχει περισσότερη εναρμόνιση και είναι πιο αποτελεσματική η αναπτυξιακή βοήθεια. Με το που θα αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και θα, δεν θα βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κουμπαράς της Ένωσης θα μικρύνει. Το θέμα είναι τι θα κάνει τα χρήματα που δίνει τώρα η Βρετανία, μπορεί να τα βάλει αλλού σε άλλες πλατφόρμες πολύπλευρες, πολυμερείς και αυτό που ίσως οδηγήσει το οποίο είναι αρνητικό σε περισσότερη κατάτμιση. Είναι αρκετά τα ποσά για να κάνουν τη διαφορά. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και όσο περισσότερο αυξάνουμε τη συνεργασία τότε έχουμε καλύτερο μείγμα πολιτικής η αναρμόνιση, η συμπληρωματικότητα, οπότε αυτά είναι ένα φρένο στις αρνητικές συνέπειες. Τώρα για να δούμε κάποιες πρακτικέ πρακτικές ε, σκέψεις, είναι νομίζω σαφές, μιλώντας σε αξιωματούχους της Ένωσης, θα συνεχιστεί η συνεργασία. Δεν μπορεί να σταματήσει η συνεργασία. Ιδίως σε επίπεδο χώρα. Φυσικό του τρόπο θα συνεχιστεί η συνεργασία. Εκεί οι επίσημε συμφωνίε είναι λιγότερο σημαντικές μέσα από τις πρεσβείες της Βρετανίας. Ε, ο συνομιλητής θα είναι η τοπική κυβέρνηση κάθε φορά για συγκεκριμένους τομείς, οπότε και νομίζω ότι εκεί θα συνεχιστεί ανεμπόδιστα η συνεργασία. Σε άλλα όμως επίπεδα για τη διαμόρφωση της πολιτικής ας πούμε θα πρέπει να επιδειχθεί ευελιξία. Θα αλλάξουν βέβαια οι όροι και προϋποθέσεις αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Ζητεί κάποια πράγματα θα ένα βασίλειο και προσφέρει κάποια άλλα. Υπάρχουν μηνύματα συνεργασία. Σα παραπέμπω στο non-paper. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει ε, ε, πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίω όσο προχωράει η υπόθεση του MFF, και θα έχει σημασία η κάθε πλευρά πόσο στρατηγικό έλεγχο θα μπορεί να ασκεί. Θα δούμε τι θα γίνει με τα καταπιστεύματα, τι υπάρχει και τι έχει στον προπολογισμό, τι θα γίνει τώρα με το EDF θα μπει στον προπολογισμό, τι θα γίνει με την διευκόλυνση, με το όργανο ειρήνευσης. Και εδώ θα χρειαστεί στρατηγικό διάλογο και συνεργασία. συνεργασία σε σχέση με τον προπολισμό είναι πιο δύσκολη και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ελπίζω ότι θα μπει και αυτός διαμορφεύσει όμως, δεν θα το εξαιρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε με τι τρόπους ε, κάποια ταμεία, κάποιοι πόροι ε, ε, θα καλυφθούν. Όλα αυτά πρέπει να ζητηθούν και να μην βγουν από τις διαπραγματεύσεις. Οπότε σε αυτή τη φάση του MFF το κλειδί είναι να αφήσουμε την κάθε πόρτα, κάθε δυνατότητα ανοιχτή. Να υπάρχουν επιλογές. Προσοχή, μην κλείνουμε καμία πόρτα. Είναι κατακλείδη, επομένω έχω αναφέρω τα εξή δύο. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει στην συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, και σας είπα κάποιους τομείς που αυτό είναι σημαντικό και αν η συνεργασία μπορεί να γίνει μόνο εκτός προϋπολογισμού και δεν ε, ε, είναι ξέρω, και συνεργασία για τον προϋπολογισμό αλλά τέλος πάντων εάν υπάρχει τέτοια συνεργασία αυτό είναι και το καλύτερο σενάριο τόσο ώστε να υπάρχει διαθεμψιακή συνεργασία έστω και εκτός του προϋπολογισμού. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτή η πόρτα για στενή συνεργασία και να εξασφαλιστεί ότι στο MFF θα υπάρχει δυνατότητα στην Συμφωνία Αποχώρησης να υπάρχει μια διάταξη ευρεία που να καλύπτει τη δυνατότητα, την πιθανότητα συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου θα χρησιμοποιήσω και το ίδιο που είπα για τις ε, λιγότερο αναπτυσσμένες χώρες. Εδώ η έμφαση έχει δοθεί και στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή, οπότε παίρνουμε χρηματοδότηση και την ε, διαθέτουμε αλλού. Η Claire Godfrey τώρα θα λάβει το λόγο, είναι μέλος της Concord Ηνωμένου Βασιλείου, έχει κάνει πολλή δουλειά ε, στην ανάλυση των επιπτώσεων του Brexit. Claire, λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν παίρνουμε πολλές ευκαιρίες για να το κάνουμε, είναι αλήθεια, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Η πλατφόρμα μας είναι μια πλατφόρμα αναπτυξιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό λοιπόν υπαγόμαστε όλοι στην Concord. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω πάνω σε αυτά που ανέφερε ο James, τα οποία φυσικά έχουν άμεση σχέση με αυτά που θέλω να πω εγώ. Είναι μάλιστα συμπληρωματικά, ε, διότι δίνουν το γενικότερο πλαίσιο. Θα σας μιλήσω από την ε, οπτική γωνία της κοινωνίας των πολιτών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Έχουμε ανοίξει διάλογο με τα μέλη μας έτσι ώστε να μάθουμε τι ακριβώς θέλουν από το Brexit, ποια θα θέλουν να είναι τα αποτελέσματα και τι πρέπει να περιμένει η κοινωνία των πολιτών από αυτό. Εντοπίσαμε τέσσερις βασικούς τομείς. Ο πρώτος από αυτούς, και αυτό έχει άμεση σχέση με ε, όσα μας είπε ο Τζέιμς, είναι η συνεχιζόμενη συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουν τη συνεργασία σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς και σε επίπεδο προγραμμάτων που πρέπει να συνεχιστούν, κοινό προγραμματισμό και σε επίπεδο πολιτικής με διεθνή συνεργασία εν ώψη των εξελίξεων και με κοινό θεματολόγιο, διεθνές θεματολόγιο το οποίο θα υπερασπιζόμαστε από κοινού σε διεθνή φόρα. Διότι πιστεύουμε ότι η συνεργασία θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Τώρα, σε ορισμένα, σημεία, σε ορισμένα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου η ανάπτυξη υπάγεται στη νομοθεσία περί ανάπτυξης, υπάρχουν προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικά ε, δεσμευόμαστε από τις σχετικές συνθήκες που έχουμε υπογράψει και από την συνένεση για την ανάπτυξη. Φυσικά η συνεργασία δίνει τη δυνατότητα τόσο στον Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν παγκόσμιο ε, αντίκτυπο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και όπως είπε και ο Τζέιμς θέλουμε να διερευνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες με ευέλικτα μέσα που θα επιτρέπουν τη συνεργασία και σε δημοσιονομικό το οποίο θα διέπεται από πρότυπα και στόχους δεσμευτικούς. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας της ε, συνέχισης, δηλαδή της συνεργασίας. Τώρα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το ζητούμενο είναι να έχει ωφέλη ε, για τους ε, φτωχότερους και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Αυτό γιατί η βοήθεια, το εμπόριο, οι επενδύσεις, ε, χρηματοοικονομικά και περιβάλλον είναι τομείς όπου θα αλλάξουν τα δεδομένα Και φυσικά, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ιτημένος θα είναι ο πιο φτωχός στις πιο φτωχές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί η καλή συνεργασία. Μία ακόμα κατευθυντήρια γραμμή είναι να μεταφερθούν όλες οι διεθνείς συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε σε επίπεδο ένωσης στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και ό,τι δεν αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξεταστεί. Για παράδειγμα, η διάσκεψη για την επισητιστική βοήθεια είναι ένα μόνο από τα παραδείγματα. Αυτές είναι οι τρεις από τις τέσσερις βασικές αρχές που διαπούν το έργο μας. Θα περάσω στην τέταρτη σε λίγο. Να πω πριν ότι όπως ε, είπα νωρίτερα, δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα είναι οι εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε ένα μακροσκελέστατο non-paper, το οποίο προσπαθεί να διερευνήσει τους ε, πιθανούς τρόπους με τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει ε, την συνεργασία μια συνεργασία που θα είναι ως το δυνατόν στενότερη για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, για, της για το κλίμα, κτλ. Η... Στην κοινή επιτροπή ε, επανέλαβε ο Υπουργός μας αυτά που έχετε ήδη ακούσει και είχε μάλιστα αρκετά θετική άποψη για την έκβαση της, ε, των συνομιλιών. Τώρα, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει σε ένα προσχέδιο για τις διαπραγματεύσεις, το οποίο όμως δεν αναφέρεται στην συνεργασία. Φυσικά αυτό είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης, γι' αυτό και δεν γνωρίζω ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσημα τουλάχιστον. Επίσης, οι απειλές νομίζω πως θα παραμείνουν και μετά το Brexit και ανεξάρτητα από αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά από τώρα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της ε, βοήθειας και της ανάπτυξης ε, με την ε, ασφάλεια. Ούτε από την πλευρά του Εμένου Βασιλείου, ούτε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περασμένη εβδομάδα η Πρωθυπουργός υπέβαλε μια πρόταση για συνεργασία και εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει διάφορα μέσα ε, που θα διασφαλίσουν την ε, συνέχιση του θεματολογίου για την ασφάλεια. Αυτό είναι κάπως ανησυχητικό. Παράλληλα, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στέλνει παρόμοια μηνύματα με την αυξανόμενη ευελιξία, με προϋπολογισμό που θα μπορεί να κατευθυνθεί πολύ εύκολα προς, ε, ανά, προς ανάγκες ε, που θα προκύψουν σε θέματα ασφάλειας, για παράδειγμα. Επίσης υπάρχει το θέμα του ε, επαναπατρισμού των κονδυλίων, αν θέλετε. Αν τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή εάν θα επενδυθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα εταιρική σχέσης. Τέλος, περνάω στην τελευταία αρχή, το τελευταίο κεντρικό θέμα που αφορά την κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό η κοινωνία των πολιτών να έχει φωνή, τη δική της φωνή, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ε, γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις ε, αντίστοιχες οργανώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε ακόμα κάποια ε, επαφή και ελπίζω να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία εταιρική σχέση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνία των πολιτών να συνεισφέρει με εμπειρογνωμοσύνη, με γνώση, με εμπειρία στις διαπραγματεύσεις. Ένας άλλος τομέας αφορά τις επιπτώσεις της συνεργασίας μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δίνει μεγάλη έμφαση στην ε, ανάπτυξη, στην ε, πρόσπιση των δικαιωμάτων στα διεθνή φόρα, μοιραζόμαστε τις απόψεις για την ε, οικοδόμηση ικανοτήτων και φυσικά μην ξεχνάμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο δυναμικό για τη διοργάνωση εκστρατιών, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Σε γενικές γραμμές λοιπόν θα υπάρχουν απώλειες στον τομέα αυτών εάν ε, κόψουμε τους εδεσμούς που μας ενώνουν. Χρειάζεται αντίθετα να ενταθεί η συνεργασία μας μετά το Brexit έτσι ώστε να μην χαθεί το δυναμικό αυτό. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή επικρατεί μια γενικότερη σύγχυση για τη χρηματοδότηση των μη κυβερνικών οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα από την ε, κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχει μια ρήτρα στις συμβάσεις με τις βρετανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις η οποία περιέχει μια περίπτωση όπου θα αποσυρθεί η χρηματοδότηση αν ε, οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο ή αν ε, αποτύχουν. Ακριβώς επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συνεισφέρει πλέον στον προϋπολογισμό. Υπάρχει όμως ε, κάποια σύγχυση και εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι βλέπουμε από τους διάφορους εράνους που γίνονται ότι αυτό ερμηνεύεται ως ε, διακριτική μεταχείριση εις βάρος ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν θα είναι σε θέση πλέον να λαμβάνουν χρηματοδότηση να κερδίζουν διαγωνισμούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανεπίλητο θέμα που επήγει. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τις μη κυβερνητικέ οργανώσει. Γνωρίζω ότι είστε μέλο τη Concord, αλλά δεν γνωρίζω αν βρετανικέ ε, ΜΚΟ, οι μεγάλε τέλο πάντων, αν έχουν γραφεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Concord, α πούμε, είναι ανοιχτή σε σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ε, απαντήστε μου σε αυτό πρώτα και τις υπόλοιπες αργότερα. Μάλιστα. Η Concord είναι ανοιχτή σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να είναι μέλος της Concord. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία διότι σε ορισμένου τομεί η, συνεργασία αυτή ξεπερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι συμβαίνει εκεί. Φυσικά οι διάφορες ε, ομάδες οργανώσεων θα συνεχίσουν τη συνεργασία όπως πριν. Ίσως ε, νομίζω πως θα υπάρξει μια ανακατάταξη σε ό,τι φορά το ποιο ηγείται ποιων προγραμμάτων, ακριβώς γιατί ορισμένες βρετανικές ΜΚΟ είχαν ηγετικό ρόλο λόγω του μεγέθους τους. Ίσως λοιπόν αυτό θα αλλάξει εις βάρος των Βρετανικών ΜΚΟ. Θα συνεχίσει όμως η συνεργασία ε, με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, ε, James έχω την ίδια άποψη για τα βασικά θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να πείτε ε, δύο λόγια για τις ε, επιπτώσεις ε, στην πράξη. Τι γίνεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα αλλάξουν. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια ένδειξη από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το αν επιθυμεί να συνεχίσει το συντονισμό σε ορισμένες περιπτώσεις. Έπειτα δεν αναφέρθηκαμε καθόλου στη Συμφωνία του Κοτονού. Νομίζω πως έχουν γίνει κάποια πράγματα, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ε, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και η Γαλλία, όπως και το Βέλγιο, έχουν ε, σχέσεις με αυτές τις χώρες που ε, ξεπερνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε πίσω στην απεικιοκρατία. Και αυτές οι χώρες λοιπόν δεν μπορούν να καταλάβουν και να φανταστούν τι θα συμβεί εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από αυτή τη συμφωνία. Έχετε λοιπόν κάποια πληροφορία, κάτι που μπορείτε να μας πείτε πάνω σε αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Για το πώς έχουν τα πράγματα επί τόπου θα έλεγα ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να φροντίζει να για τη συνεργασία με κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει μια το, ε, συνεργασία στο τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας. Η συνεργασία υπάρχει. Φυσικά σε κάποια ε, στιγμές η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ε, γίνεται η συζήτηση ε, και κλεισμένων των θυρών κατά κάποιο τρόπο, μόνο μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν συμφωνίες για δημοσιονομική υποστήριξη και αυτό το μοντέλο λειτουργεί αρκετά φυσικά θα έλεγα πρόσφατα. Συμμετείχαμε ε, στην αξιολόγηση του μηχανισμού για την ειρήνη στην ε, Αφρική. Ε, υπάρχει σημαντική υποστήριξη για τους στόχους αυτούς του μηχανισμού, του μηχανισμού υπάρχει θέληση να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πώς θα γίνει ακριβώς παραμένει ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά πάντως το μηχανισμό για την ειρήνη στην Αφρική, είναι πολύ σημαντικό να αναζητηθούν ε, δύο συνεργασίας, ε, γιατί, ε, για παράδειγμα, η Γαλλία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτό το τομέα και χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη. Αυτά για την Αφρική και ε, υπάρχει συνεργασία και με την ε, Αφρικανική Ένωση και είναι πολύ σημαντική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. ό,τι αφορά τη Συμφωνία του Κοτονού, κατά κάποιο τρόπο ανοίγουν νέες ε, δυνατότητες, γιατί αυτή η συμφωνία δεν είναι μέρος κάποιων διεθνών συνθήκων. Νέα κράτη από την Αφρική Καραϊβική και από τον Ειρηνικό έχουν ε, υπογράψει τη συμφωνία. Ίσως ε, κάποια άλλα θα ε, τολμούσαν να, να το κάνουν στο μέλλον και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια ευρωπαϊκή συνεργασία με ε, τις χώρες της Αφρικής, ε, της Καρυβικής και του Ειρηνικού, με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Φυσικά χρειάζεται πολύ σκέψη για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Προλά κράτη-μέλη θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές της συνεργασίας και ε, με τις χώρες Αφρικής, ε, Καραβιακής και του Ειρηνικού. Δεν είναι πρώτη φορά που προτείνεται η εγγραφή στον προϋπολογισμό ε, συγκεκριμένων ε, δράσεων σε αυτές τις χώρες. Ε, ίσως θα ήταν καλό να μην εγγραφούν στον προπολογισμό κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε τη δυνατότητα στενής συνεργασίας ανάμεσα ταυτόχρονης χρήσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και από άλλες πηγές. Αν η ευρωπαϊκοί θεσμοί και κυρίως τα κράτη-μέλη που ε, υπογράφουν τη συμφωνία θα μπορούσαν μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο να φανταστούν ε, λύσεις για να συνεργαστούν στα πλαίσια της συμφωνίας του Κοτονού. Πρέπει να έχουμε φαντασία ε, φυσικά και χρειάζεται πολιτική βούληση. Και πρέπει επίσης η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να καθορίσει ακριβώς τι θέλει. Δεν βλέπω κάποιος άλλος να θέλει να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, παρουσιάσεις. Σίγουρα θα ξανασυναντηθούμε και θα συζητήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ και πάλι.

Συνάδελφοι, περνάμε στο τελευταίο σημείο τη σημερινή διάταξη, το σημείο 14 για σήμερα. Ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη μειώνοντα τη φτώχεια μέσω τη τεχνολογία. Συμφωνήσαμε να συντάξουμε μία έκθεση πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα. Γι' αυτό καλέσαμε και κάποιους εμπειρογνώμονες. Η συγητής είναι ο Μπόγναν για αυτή την έκθεση. Συναντηθήκαμε και ε, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγάντα είδαμε την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Κάποιοι συμμετέχουν σε ε, προγράμματα κατάρτισης ε, εικονικής πραγματικότητας. Ε, και νέοι ε, συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ε, σχετικά με τις ψυχιακές τεχνολογίες. Γνωρίζουμε όλοι τον αντίκτυπο της χρήσης των κινητών τηλεφώνων σε αναπτυσσόμενες χώρες τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα. Σήμερα ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ε, Αφρικής χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα και το σήμα πολλές φορές είναι καλύτερο από ό,τι στο κέντρο του Λονδίνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση, ε, μέσα από το καταπιστευματικό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αφρικής που ιδρύθηκε το 2007 καθώς και μέσα από το Μηχανισμό Συνεργασίας για την Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ε, σήμερα έχουμε ε, εκπροσώπους από την GIZ και από την EMEA Satellite Operators Association. Θα ήθελα πολύ να μου εξηγήσετε τι σημαίνει το ακρόνιμο EMEA και είναι εδώ επίσης ο κύριος Μπόντο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος θα μιλήσει για το τι κάνει η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ πάνω σε αυτά τα θέματα. Πρώτο έχει το λόγο ο κύριος Ρίχτερ. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων χωρίς έγγραφο εργασίας γιατί πρέπει να εντοπίσουμε τους τομείς όπου θα είναι μεγαλύτερος αντίκτυπος. Θα συζητήσουμε για παράδειγμα το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη. Ε, υπάρχουν περιορισμοί, άρα πρέπει να ορίσουμε τους τομείς στους οποίους ο αντίκτυπος θα είναι ε, μεγαλύτερος. Κύριε Ρίχτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να μιλήσω εδώ σήμερα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το D4D ε, σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο μετά από τη συμμετοχή μας σε συναντήσεις πέρσι και τις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο. Υπάρχουν επαφές και συνεργασίες σχετικά με την ψηφιοποίηση και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ένα στρατηγικό έγγραφο στη Γερμανία για την ψηφιακή ανάπτυξη ε, που ε, ορίζει ως στόχο μια ψηφιακή επανάσταση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το μέλλον μας είναι ψηφιακό. Υπάρχουν τρόποι να καταστεί η διαδικασία πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν πολλά ε, παραδείγματα διαφορετικών δράσεων. Είναι νέο αυτό το ζήτημα. Ε, η ε, Γερμανική Υπηρεσία Συνεργασίας προσπαθεί να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους ε, οι δράσεις θα είναι πιο αποτελεσματικές και θα ε, αξιοποιηθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο οι ψηφιακές τεχνολογίες, η καινοτομία, δημοκρατία, ε, πρόσφυγες φυσικά στην καρδιά όλων αυτών των ζητημάτων βρίσκονται η απασχόληση βρίσκεται η απασχόληση η ψηφιο επίση ε, υποστορίζεται όλο ένα και περισσότερο και συζητείται ε, στη Γερμανία. Η οικονομική ανάπτυξη, η χρηστή διακυβέρνηση, η υγεία και η εκπαίδευση είναι οι τομείς ε, ε, με τις καλύτερες προοπτικές. υπάρχουν εταίροι που ε, ζητούν την ένταξη των ψηφιακών ε, τεχνολογιών στις δράσεις. Χρειάζονται συστήματα διαχείρισης των ψηφιακών γνώσεων, ε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της διαχείρισης των δεδομένων και στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται ε, συστήματα διαχείρισης των big ε, data μεταξύ άλλων, προκειμένου να υποστηριχτεί και η συνεργασία για την ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες ε, πρωτοβουλίες σε αυτούς τους διάφορους τομείς και οι εμπειρογνώμονες ζητούν περισσότερη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων. Ξέρουμε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες ε, πρέπει να ε, αξιοποιηθούν στα πλαίσια συγκεκριμένων ε, σχεδίων και δράσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια των συνεργασιών και φυσικά αντλούμε διδάγματα. Από τις Επιτυχίες είναι η πρωτοβουλία του G20 για την απασχόληση. Υπάρχει μια δέσμευση ε, του G20 προκειμένου να ε, ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών και των ε, κοριτσιών με πρωτοβουλία της Γερμανίας. Υπάρχει και πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των καλύτερων ιδεών ε, για την ε, συμμετοχή ε, γυναικών και κοριτσιών στις διάφορες δράσεις. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με την UNESCO για τη διαμόρφωση μιας εργαλειοθήκης για την καλύτερη συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και ε, ε, σχετικά με συστήματα υποστήριξης των ε, startups. Και υπάρχει το θέμα της τεχνικής υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης. Σε συνεργασία με τα μέλη του G20 πρόκειται για ένα πρωτοκόλλο που υπογράφηκε πέρσι, υλοποιείται ήδη επιτόπου ε, σε διάφορα ε, σχέδια και στα πλαίσια διάφορων δράσεων, σε ε, εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Φέτος έχουμε δράσει στην Νότια Αφρική και στη Μοζαμβίκη μεταξύ άλλων. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των νεοφιών επιχειρήσεων, πιστεύουμε ότι πρέπει να υποστηριχτούν οι ψηφιακές startups και να υποστηριχτεί και η παροχή υπηρεσιών. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν διάφορες συνεργασίες με επιχειρήσεις, Orange, IBL, μεταξύ άλλων, αλλά και με παρόχους ε, χώρων ε, κοινών χώρων ε, εργασίας στην Νότια Αφρική. Και στην Κένια και στην Ιγυρία ε, υλοποιούνται ε, δράσεις και στην Τινησία και στην Κάνα. Στόχος είναι να υποστηριχτούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και γενικώ το, όλο το οικοσύστημα αυτών των επιχειρήσεων που ε, δημιουργεί καινοτομία και αξιοποιεί κεφάλαια, δημιουργεί ε, απασχόληση επιτόπου. Ο πρόεδρος της Νιγηρίας ε, ζήτησε ε, την συμβουλή μας για την υποστήριξη ενός βιώσιμου συστήματος βοήθειας στις startups και πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για ένα βιώσιμο σύστημα νεοφιών επιχειρήσεων. Υπάρχουν ιδέες και στο τομέα της υγείας. Υποστηρίζουμε στη Δυτική Αφρική ε, συστήματα αντιμετώπισης των ε, πανδημιών. Σε περίπτωση πανδημίας στη Δυτική Αφρική στόχος είναι να δοθεί μια βιώσιμη ε, απάντηση και να αξιοποιηθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση του κοινού. Αυτή η δράση ε, υλοποιείται και ε, σε άλλες περιοχές. Η συζήτηση για την ψηφιοποίηση αφορά πολύ συχνά και τα drones. Αυτή η συζήτηση όμως είναι πολύ τεχνική συχνά. Τι μπορούν να υποστηρίξουν τα drones. Ε, μια ιδέα υπάρχει στην Τανζανία για την παράδοση φαρμακευτικών προϊόντων σε στην Ήπεθρο. και συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Τανζανίας για την υλοποίηση αυτού του ε, σχεδίου προκειμένου να ε, υπάρχει, να επιτευχθεί στοχευμένη παράδοση φαρμάκων στην Ήπεθρο ε, στόχος είναι να γίνει κάτι τέτοιο δυνατό και σε περιοχές που πλήττονται από ε, συγκρούσεις. Στη Ρουάντα η κυβέρνηση ε, υποστηρίζει την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου διευκολυνθεί η χρήση των drones Και τώρα ε, τα drones χρησιμοποιούνται και στην ε, Ρουάντα στα πλαίσια ε, δράσεων συνεργασίας για την ανάπτυξη μαζί με διάφορους εταίρους. Υπάρχουν παράλληλα και πρωτοβουλίες της Αφρικανικής Ένωσης που υλοποιούνται ταυτόχρονα με τις δικές μας στο τομέα της ανάπτυξης Συνάδελφοι μόλις επέστρεψαν από μια ε, αφρικανική διάσκεψη στο τομέα της ανάπτυξης. Υπάρχει και το θέμα της χρήσης ε, συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ε, υλοποιούνται σχετικές δράσεις ε, και στο Μπαγκλαντές μεταξύ άλλων προκειμένου να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στα συστήματα ελέγχου της δικαιοσύνης Αυτό ε, αφορά διάφορα ε, θέματα. Στο Μπαγκλαντές πρόκειται απλώς για παραδείγματα ε, σε συζητήσεις με την κυβέρνηση, με υπουργούς και πολιτικούς προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες. Θα έλεγα ότι σε πέντε χρόνια ε, μάθαμε ότι χρειάζονται νέε συνέργειες με επιχειρηματίες, με κυβερνήσεις. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται νέες μορφές ε, συνεργασίες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, χρησιμοποιούμε τις παλιές μορφές συνεργασίες για την ανάπτυξη όσο έχει. Υπάρχουν νέες ε, ομάδες ε, τις οποίες ε, στοχεύουμε. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζονται ικανότητες, χρειάζονται πόροι όμως για την υπολοποίηση των λύσεων. Πολύ συχνά περιοριζόμαστε σε συζητήσεις που αφορούν την Κένια, την Ιγυρία... Ε, στην, στην Ήπεθρο υπάρχουν όμως πολύ μεγαλύτερες προπτικές από ό,τι φαντάζεστε. Υπάρχει το θέμα των ε, ψηφιακών σχεδίων. Έχω πάει ο ίδιος στο Πακιστάν πριν από ένα χρόνο. Το Πακιστάν δεν θέλει να θεωρηθεί ε, ε, ως αδύναμη ε, χώρα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Φροντίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να αντλήσει διδάγματα. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση γιατί οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν περιορίζονται από σύνορα. Στο μέλλον η απάντηση της GIZ ποια είναι. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε σχέδια για την αξιοποίηση τεχνολογιών τύπου blockchain. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν κάποιες ε, τάσεις, αλλά ε, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι μπορεί να ε, αξιοποιηθεί στη πράξη στο τομέα των τεχνολογιών blockchains. Προσπαθούμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες σύναψης νέων συμφωνιών συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το σύστημα συνεργασίας και δεν πρέπει να παραμελήσουμε καμία διάσταση. Υπάρχει καινούριο προσωπικό στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις ψηφιακές τεχνολογίες και δημιουργούνται νέες ε, υπηρεσίες. Και αυτό που ενδιαφέρει στη σημερινή συζήτηση είναι η απόφαση να χρησιμοποιηθεί να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές ε, τεχνολογίες, γιατί το, ε, στην πράξη πραγματικά, γιατί το θέμα δεν είναι αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά να χρησιμοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα εργαλεία και αν κάποιος δεν χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία πρέπει να το δικαιολογήσει. Αυτό είναι κάτι καινούριο για το τομέα της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη στη συνεργασία. Ε, για μας οι ε, ψηφιακές τεχνολογίες είναι το μέλλον και ήδη οι εταίροι μας ζητούν την αξιοποίησή τους. Και αυτό σημαίνει ότι ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η, η, διάσταση για, στα πλαίσια της ορπίσης των 2.000 ε, δράσεων που υλοποιεί η GIZ ε, και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω... Ε, έχω μια ερώτηση. Αυτό το blockchain που είπατε, τι σημαίνει ακριβώς, δεν, δεν ξέρω. Είναι μια τεχνολογία όπως αυτή που χρησιμοποιεί η Fintech για παράδειγμα η οποία χρησιμεύει για να αξιολογηθεί το δυναμικό της τεχνολογίας. Είναι μια τεχνολογία δηλαδή η οποία αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες σε διάφορους ε, υπολογιστές οι οποίες πληροφορίες μπορούν να εντοπιστούν. Το υλικό δηλαδή αυτό ε, είναι δυνατόν να ιχνηλατηθεί και να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι το blockchain. Έχει συζητηθεί και στο πλαίσιο της ΤΕΠ e και έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα, διότι θεωρητικά τουλάχιστον μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ανήκει να έχει τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να χρειαστεί να πάει να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή, ένα πολίτη στην Τανζανία μπορεί να έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό στο κινητό τηλέφωνο. Τώρα, το πώ θα φτάσουμε μέχρι εκεί, αυτό είναι ε, κάτι που θα καθορίσει το πόσο καλά θα χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι αρκετά τεχνικό θέμα, πρέπει να υλοποιηθούν πολλά επιμέρους ε, πράγματα, όμως θα είναι ένα τεράστιο άλμα για την ε, τεχνολογία. Μάλιστα, δεν είμαι σίγουρη αν το κατάλαβα, ωστόσο. Δηλαδή, είναι ας πούμε, είναι μία ε, πρόταση π.χ. για το πώς θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στη Γεωργία. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι δικαστικές αποφάσεις αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με το blockchain θα δώσεις τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στοιχεία τα οποία δεν θα μπορούν να διαγραφούν. Δηλαδή, δημιουργείς έναν ε, ηλεκτρονικό εγκέφαλο, ας πούμε, μια συλλογική μνήμη σε διάφορα τερματικά. Η πληροφορία αυτή δεν μπορεί ούτε να διαγραφεί, ούτε να ε, τροποποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν ε, η χνηλασιμότητα. Για παράδειγμα, το κτηματολόγιο στη Λατινική Αμερική. Η Αργεντινή έχει εισαγάγει ένα σύστημα όπου ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο και αν κάποιος αλλάξει κάτι μπορούν αυτό ταυτόχρονα να το δουν όλοι και να δουν τι έχει αλλάξει και γιατί. Είναι ένα σύστημα που δίνει περισσότερη διαφάνεια. Χρησιμοποιείται δηλαδή η τεχνολογία για να ε, βελτιώσει τη διαφάνεια. Είναι στην ουσία ένα εργαλείο το οποίο ακόμα ε, ψάχνουμε να βρούμε την ε, προστιθέμενη αξία του. Ψάχνουμε να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε με την τεχνολογία να βελτιώσουμε το μέλλον και επειδή ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ερευνές μας για τη χρήση του, ακόμα τα αποτελέσματα κρεμούν. Έχουμε αρκετό δρόμο λοιπόν ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο μιλητή, την κυρία Χόλα, από τη Γενική Γραμματεία της, ε, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μέσης Ανατολής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Βέντα. Είμαστε ένα σύνδεσμος οργανώσεων που ασχολούνται με τις δορυφορικές επικοινωνίες Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Παρέχουμε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο και θα ήθελα να σημειώσω για όσους βρίσκονται εδώ ότι οι ε, πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις ε, δορυφορικών τηλεπικοινωνιών εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα και λοιπόν έχετε επιχειρήσεις και στην Αφρική κάτι που φυσικά έχει σχέση με αυτά που λέμε τώρα. Ναι, αυτό που κάνουμε είναι να συνεργαζόμαστε με διάφορους ε, ηθήνοντες χαράξεις πολιτικής έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξελίξεις της τεχνολογίας έτσι ώστε η χάραξη πολιτικής να προκύπτει μετά από ενημερωμένες... Ε, μετά από ενημέρωση. Βλέπουμε πως υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Ο κόσμος υποφέρει, γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε την δορυφορική τεχνολογία. Τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ο κυριότερος λόγος γι' αυτό είναι η έλλειψη υποδομών τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι και η αιτία των προβλημάτων σε κάθε μέρος του κόσμου. Τώρα, πώς μπορεί να βοηθήσει το διάστημα. Ένας δορυφόρος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο 1 τρίτο της ε, επιφάνειας της γης. Αυτό επιφέρει και πλεονεκτήματα. Οι δορυφορικέ επικοινωνίες ε, δηλαδή δεν κάνουν διακρίσεις. Αν κάποιο ζει σε ένα απομονωμένο νησί, σε ένα βουνό, σε μια απομονωμένη, απομακρυσμένη περιοχή, το κόστος σύνδεσης αυτού του ενός ανθρώπου ε, δεν είναι υψηλότερο από εκείνο τη σύνδεση ενός ε, ανθρώπου που κατοικεί σε μια πυκνοκατοικημένη πόλη. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι δορυφορικό πιάτο, ένα δέκτη δηλαδή, και ένα ε, μόντεμ που θα συνδέεται με το δέκτη. Είναι μία λύση προφανής θα έλεγα η οποία ναι μεν συνδέει τους ε, ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα όμως επειδή δεν φαίνεται από τη γη, βρίσκεται στο διάστημα ο κόσμος δεν γνωρίζει ε, τα ωφέλη της. Μάλιστα, οι δορυφορικές επικοινωνίες ε, χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε δει δραματική πρόοδο της τεχνολογίας και αυτό φαίνεται και στις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας δορυφόρος. Τρεις μόνο έχω φέρει μαζί μου με τρεις φωτογραφίες για να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς ε, οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες κάνουν τη διαφορά. Η μία έχει να κάνει με χρηματοοικονομικά, με την χρηματοπιστωτική ύπαρξη ενός ατόμου μέσω των ε, δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Πώς μπορούμε δηλαδή μέσω δορυφόρου να υποστηρίξουμε το τραπεζικό σύστημα και να παρέχουμε υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες ε, σε όλο τον κόσμο. Ακόμα δηλαδή και σε μια βουνοκορφή και σε ένα απομακρυσμένο νησί και τα λοιπά. Ο καθένας θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα με ένα κινητό και δορυφορικά να κάνει τραπεζικές συναλλαγές. Αυτό βλέπουμε ότι βοηθά ιδιαίτερα στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες όπου προς το παρόν υπάρχουν υπηρεσίες όπως η Western Union. Μετά, αυτή η εικόνα που βλέπετε δείχνει ένα πλωτό νοσοκομείο το οποίο έχει δορυφορική σύνδεση. Είναι στο Μπαγκλαντές, είναι ένα πλοίο δηλαδή το οποίο πλέει ε, στο Μπαγκλαντές και ο κάθε μπορεί να ανέβει σε αυτό το πλοίο για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να δει ένα γιατρό και ακόμα να κάνει και μερικές μικρές εγχειρήσεις. Οι γιατροί και το προσωπικό του νοσοκομείου μπορούν μέσω της δορυφορικής επικοινωνίας να συνδεθούν με διεθνή νοσοκομεία ή και με την πρωτεύουσα της χώρας ανάλογα με το που βρίσκονται και να ε, στείλουν τις πληροφορίες των ασθενών. Οι κοινότητες τις οποίες εξυπηρετεί αυτό το πλωτό νοσοκομείο είναι κοινότητες οι οποίες ε, μπορεί να περά, στις οποίες μπορεί να ζήσει κάποιος χωρίς ούτε μία φορά στη ζωή του να έχει τη δυνατότητα να πάει σε νοσοκομείο βελτιώνει επομένω την ποιότητα ζωής. Το πλοίο αυτό πηγαίνει σε διάφορα νησιά, επιστρέφει, ε, είναι συνεχόμενο το ταξίδι του, δεν υπάρχει κάποια διακοπή των υπηρεσιών, το οποίο είναι καλό. Υπάρχει μια πλατφόρμα με το όνομα SatMed, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά και στην Ασία και στην Αφρική. Τέλος, κινητή συνδεσιμότητα. Όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι τεράστιο το δυναμικό που έχει ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δώσει σε κάποιον, του βάλει στο χέρι ένα κινητό τηλέφωνο, δεν ξέρει πώ μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ένα αγρότη μπορεί να κοιτάξει τι τιμέ των ε, ε, σιτηρών, α πούμε, να συνδέσει απομακρυσμένε περιοχέ. Για να γίνει όμω αυτό, να μπορεί να συνδέσει απομακρυσμένε περιοχέ, πρέπει να χτίσει διάφορους πύργους που θα συνδέουν τις περιοχές ή να σκεφτείς ε, να το κάνεις αυτό μέσω της δορυφορικής σύνδεσης. Εδώ βλέπουμε την ε, τεράστια διαφορά, το όφελος που έχει η δορυφορική σύνδεση σε απομονωμένα μέρη όπως ορισμένα της Αφρικής. Εδώ λοιπόν ο χειριστής του δορυφόρου έχει εγκαταστήσει το δέκτη, έχει δημιουργήσει τον ε, σταθμό, χρειάζεται βέβαια ηλεκτροδότηση με φωτοβολταϊκά, οπότε πρέπει να εγκατασταθούν και αυτά και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή έτσι ώστε τα φωτοβολταϊκά που θα εγκατασταθούν να είναι βιώσιμα και να μπορούν να συντηρηθούν. Δεξιά βλέπετε το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε με δορυφορική σύνδεση στο Κονγκό, και αμέσως, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, ε, ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει ε, σύνθεση 3G από το μηδέν. Όμως, το ζητούμενο εδώ είναι πώς όλη αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερη κλίμακα και να γίνει βιώσιμη. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα. Αυτό δεν θα γίνει μόνο του. Χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις. Η πιο σημαντική θεωρώ είναι να ξεπεράσουμε την έλλειψη πληροφόρησης. Πρέπει να γίνει ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Όπως σας είπα, η δορυφορική σύνδεση είναι αόρατη, αλλά υπάρχουν και άλλα. Το Y-Gig, για παράδειγμα, έχετε ακούσει όλοι για το Wi-Fi, όμως το Y-Gig είναι η επόμενη γενιά, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους ε, ανθρώπους να αποκτήσουν ε, δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων gigabyte σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Ξέρετε πώς ε, πάει αυτό και αυτό ισχύει και για τους δορυφόρους, διότι δεν μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να αυξηθεί η ενημέρωση για τα ωφέλη των ε, δορυφορικών συνδέσεων, διότι διαφορετικά αν δεν υπάρξει ε, ζήτηση δεν θα αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτές οι τεχνολογίες να είναι προσβάσιμες, να είναι προσιτές οικονομικά, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που διαθέτουμε. Χωρίς λοιπόν ε, τον προσιτό χαρακτήρα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Και ακόμα και... Ακόμα και αν υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, για πολλές χώρες είναι οικονομικά απαγορευτική η ανάπτυξη τέτοιες τεχνολογίες και αυτό γίνεται μέσω διαφόρων ε, ρυθμιστικών φραγμών. Πιστεύουμε πως αυτά τα εμπόδια προκύπτουν από την έλλειψη ενημέρωσης, διότι εάν γνώριζαν όλα τα ωφέλη, τότε δεν θα επέβαλαν διάφορους ε, φραγμούς και εμπόδια στη χρήση τους. Για παράδειγμα, τα υψηλά τέλη για τη χορήγηση άδεια. Ε, αυτή τη στιγμή το ύψος ε, για την εγκατάσταση ενός δορυφορικού δέκτη είναι, το κόστος είναι απαγορευτικό. Και τι θα γίνει αν, προσπαθ... αν αυξήσεις το κόστος ε, σε μια εταιρεία είτε θα το μετακυλήσεις στον χρήστη, θα είναι πιο ακριβώς ο δέκτης δηλαδή, είτε θα βρει κάποιον άλλο τρόπο να το κάνει. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει άλλη λύση για αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Και πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις ε, ευκαιρίες που έχουμε εδώ και να μην τις αφήσουμε να πάνε χαμένες. Έπειτα η χρηματοδότηση πρέπει να είναι προσβάσιμη. Εδώ, συχνά, θεωρούμε πως υπάρχει έλλειψη υποδομών. Γι' αυτό ποια είναι η λύση, χρηματοδότηση για υποδομές. Είναι ένα λογικό συμπέρασμα. Όμως, οι δορυφορικές υποδομές υπάρχουν. Οι δορυφόροι βρίσκονται στο διάστημα ήδη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη εξετάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το παρουσιάσαμε στους επιτρόπους και τους είπαμε ότι δεν είναι μόνο οι υποδομές που χρειάζονται χρηματοδότηση, αλλά και η πρόσβαση σε αυτές. Η τεχνολογία δηλαδή της πρόσβασης, η δορυφορική τεχνολογία τι χρειάζεται, μόνο αυτό το κουτί, το μόντεμ, που είναι μερικές εκατοντάδες ευρώ και ο δέκτης. Και είναι πολύ μικρό το κόστος αν το συνδέσουμε με, αν το συγκρίνουμε μάλλον με, την, με τις κινητές ε, τηλεπικοινωνίες. Θεωρούμε πως πρέπει να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών έτσι ώστε να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα για να υλοποιήσουν στόχους προς το δημόσιο συμφέρον είτε για ηλεκτρονική μάθηση, ψηφιακή ε, ψηφιακό αλφαβατισμό, εκπαίδευση, γεωργία. Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να ε, βελτιωθεί η κατάσταση, να καλέσουμε επιχειρήσεις, ε, να ενημερωθούν, να ανταποκριθούν στις ε, ανάγκες της τοπικής τους κοινωνίας, τις οποίες μάλιστα γνωρίζουν. Τώρα, συνδεσιμότητα κινητές τηλεπικοινωνίες. Βλέπουμε εδώ ότι ότι το σύστημα έχει κατασταθεί από ντόπιου και θα συντηρηθεί από ντόπιου. Γι' αυτό αυτό μας λέει πως θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας επιτόπου. Μας ανοίγει νέες, ε, μας δίνει δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Έχουμε και επιτυχία στου αναπτυξιακούς, ε, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Προσπαθούμε λοιπόν να στο πλαίσιο του διαλόγου με διάφορες κυβερνήσεις να δούμε τις ανάγκες τους. Μας λένε ότι θέλουμε να εστιάσουμε στο δίκτυο 5G. Δεν μπορούμε να ε, γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα ή το αντίστροφο. Δεν θεωρούμε κατά ανάγκη πως αυτό είναι λάθος. Αυτές οι προτεραιότητες είναι βέβαια διαφορετικές, δεν χρειάζεται όμως να είναι και ανταγωνιστικές. Και το 5G και ε, οι καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος είναι εξίσου σημαντικές και πρέπει λοιπόν οι πολιτικές που θα σχεδιαστούν να χαρακτηρίζονται από συνέπεια τόσο σε ό,τι αφορά επενδυτική πολιτική κτλ. όσο σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Είναι μια τεράστια πρόκληση αυτή, αλλά ταυτόχρονα και τεράστια ευκαιρία που θα ωφελήσει πολλούς. Και το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί είναι η φωνή των πολιτών και κυρίως η φωνή των πολιτών που δεν μπορούμε να ακούσουμε διότι δεν είναι συνδεδεμένοι και δεν γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις που θα επηρεάσουν στη ζωή του, τη ζωή τους. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ε, λήψη αποφάσεων που θα αλλάξει το μέλλον των πολιτών αυτών. Στην Ουγγάντα είδαμε πάρα πολλά ηλιακά πάνελ Πήγε για τηλέφωνο, τηλεόραση κλπ. Μπόγκταν. Έχει την πρόβληση τη φτώχεια όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Παγκοσμίω. Θα δούμε πώ στην ε, πολιτική ανάπτυξη θα αξιοποιήσουμε την ψηφιοποίηση, ε, ανέλαβα τη σχετική και την συνεργασία. Μιλούμε πολύ για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την συνεργασία. Μιλούμε πολύ για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά ε, ακόμα έχουμε οραγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το 5G και θέματα προσβασιμότητας με το 5G, το 3G για το ίντερνετ. Οπότε δεν είχε πολύ συνάδελφοι εδώ θα, γιατί θα ήθελα να ακούσω τι έχουν να πούν οι σκιώδες ηγητές. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι. Ξέρω τους κλειμένους μας. τι γίνεται με την δημοσία υγεία, τι γίνεται με την απασχόληση. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρο. Μόνο ένα από του κύριου είναι εδώ, ο Ενρίκη Γκερέρο. Ευχαριστώ για την ε, τόσο πλήρη παρουσίαση. Και εγώ δεν κατάλαβα και τόσο καλά την υπόθεση blockchain. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Πάντως το υποσυνειδητό μου είναι αυτά για τα εικονικά νομίσματα. Πέραν αυτής της λεπτομέρειας, Μπόγκταν, έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ότι όλες πολλές πτυχές και στην συνάντηση κορυφής ένα από τα θέματα ήταν το πώς θα ληφθούν κάποια μέτρα καινοτόμα, ούτω ώστε να βοηθηθούν αυτοί που έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτά τα καινοτόμα μέτρα, σύνδεση ε, υγειονομική κάλυψη, χρηματοδότηση για το εμπόριο, ας πούμε, αντί για ανταλλαγή προϊόντων να μπορεί να πληρώσει κανείς με πιστοτική που με αυτοί που έχουν ανάγκη πεις βοήθειας επίσης ε, έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχουν ακόμα ψηφιακές τεχνολογίες. Ε, οι πρόσφυγες, κάποιοι ευάλωτοι πληθυσμοί, χώρες, αλλά όπου έχει χτυπήσει κάποια φυσική καταστροφή, κάποια θεομηνία. Οπότε θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμε οι φυσικέ τεχνολογίε. Ο ρόλο τη γυναίκα τώρα σε όλε τι μελέτε για ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης αναφέρθηκε και το μία της υγείας η αξιολόγηση του κινδύνου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για κάποιους κυκλώνες, για κάποια άλλα προβλήματα κλιματολογικά, ε, θεομηνιών, για εκρήξεις ηφαιστείων, για σεισμούς, γιατί υπάρχουν πολλά σημάδια που προηγούνται της έκρηξης, ας πούμε, του συμβάντος και σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, Μόλις δούμε την πρώτη εκδοχή του κειμένου σου θα δούμε τι θέματα μπορούμε να καλύψουμε ανθρωπιστικά και θα συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε όσο γίνεται την έκθεση. Αλλά ξεκινάει για την αντίδραση σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Δηλαδή και για απειλές από τη φύση αλλά και σε περιπτώσεις συγκρούσεων. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε με την τεχνολογία ε, πληροφορίες, σωθούν ζωές. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ρικ Μπόμ τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πόλεις, τοπικές αρχές, ψηφιοποίηση κλπ. Τα διαβάζω με τα φράσμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, πρόκειται για ένα τμήμα που ασχολείται με διάφορα ζητήματα. Σήμερα θα συζητήσουμε για την ψηφιοποίηση, αλλά ε, είναι αρμοδιότητά μας και οι πόλεις γιατί την ψηφιοποίηση και για εκεί ισχύει, ε, τοπικές αρχές επίσης και αγαπητέ κύριε Σίγητα, ε, κύριε Βέντα, αγαπητοί κύριοι ομιλητές, προσωπώ σήμερα εδώ την ντεύκο, θεωρώ θετική τη δική σας πρωτοβουλία για να έχετε αυτήν την έκθεση και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται. Να συνεργαστούμε με τον κύριο εισηγητή και επίσης εγώ και συνεργάτες και από την DG Connect. Εδώ, ο... Ξέρω, τώρα στα ισπανικά μπορώ να σας πω επίσης ότι συνεργαζόμαστε συχνά, συγγνώμη στενά με την DGECO για την ψηφιοποίηση ακριβώς για τους λόγους που εσείς κύριε Γκερέρο αναφέρατε συνεργαζόμαστε με την Γενική Διεύθυνση της ΕΚΟ και έχουμε πολλές σχετικέ σχετικές πρωτοβουλίες. Δεν έχω τα σχετικά έγγραφα αλλά σας διαβεβαιώ ότι ισχύει αυτό ότι θα βοηθήσουμε, δώσα από εμά θα βοηθήσουν και οι συναδελφοί της ΕΚΟ. Πάλι στα αγγλικά. Πρόκειται για μια ψηφιακή παράσταση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας και αυτό τώρα αντικατοπτρίζεται ως συμβολή και στην εξωτερική αγορά αλλά και στις ε, εξωτερικές πολιτικές. Και επίσης είναι καλό νέο το ότι έχει ταχεία διάδοση η ψηφιοποίηση στις χώρες μας. Και όμως ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας γιατί υπάρχει παγκόσμια μείωση των ε, συνδρομών των ευρυζωνικών αλλά ακόμα ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί στις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες και στις μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες τα πράγματα είναι ιδιαίτερως δύσκολα. Επίσης Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιφερειών της ίδιας χώρας. Διαφορά υπαίθρου πόλης όπως αναφέρθηκε και επίσης όπως αναφέρθηκε έχουμε τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών για τα ψηφιακά. Επίσης, τα οικοσυστήματα της επιχειρηματικότητας για τα ψηφιακά για διάφορους λόγους δεν προχωράνε. Είναι θέματα γλωσσικά, θέματα γραφειοκρατίας, ε, θέματα δεξιοτήτων, οπότε σας τονίζω ότι δεν είναι τώρα στο επίκεντρο της προσοχής μας τα ψυχαγά για πρώτη φορά. Τελευταία 20 ετία εμείς έχουμε προωθήσει σχετικά προγράμματα, αλλά σε βάση ad hoc. 350 εκατομμύρια ευρώ έχουν εκταμιευθεί για πρωτοβουλίες σχετικές με τα ψηφιακά τελευταία δεκαετία. Όμως, τώρα και λέει για το mainstreaming των ψηφιακών στις πολιτικές της Ένωσης προ, να χειραφετήσει ανήλικες και ανήλικες γυναίκες. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν την ζωή τα σημεία αυτού του εγγράφου τον Νοέμβριο αποτυπώθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Νοέμβριο. Η ψηφιακή υποδομή, η διακυβέρνηση, οι δεξιότητες, βοήθεια της οικονομίας και τα ε, επιχειρηματικά. Η ψηφιακή υποδομή, η διακυβέρνηση, οι δεξιότητες, βοήθεια της οικονομίας και τα ε, επιχειρηματικά οικοσυστήματα ούτως ώστε να ωφεληθούν οι μηνύα ψηλών. Βέβαια, μας ενδιαφέρει ιδίως το τι θα